είναι οι δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 29 και 30 Οκτωβρίου 2009 κλείνει η παρένθεση. Χαιρετίζω τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μπαρόζο και την κυρία Σεσίλια Μάλστρομ, που εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Καλώς ορίσατε είστε και πρώην συνάδελφός μας. Λοιπόν, δίνω το λόγο αμέσως στην κυρία Μάλστρομ, Ευρω... την Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, Βρισκόμαστε στις παραμονές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της επόμενης εβδομάδας με ένα ιδιαίτερα ε, φορτωμένο πρόγραμμα ημερήσιας διάταξης που αφορά στην ευημερία των πολιτών μας. Θα συζητήσουμε τις κλιματικές αλλαγές, θα πρέπει να βρούμε ένα δρόμο για να βγούμε από την οικονομική κρίση στην Ευρώπη, θα πρέπει να μιλήσουμε για την ενεργειακή ασφάλεια και την καταπολέμηση της ε, παράνομης ε, μετανάστευσης και όλα αυτά θα γίνουν πιο εύκολα άμα λύσουμε το πρόβλημα της συνθήκης της Λισαβόνας για να συνεχίσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις εργασίες μας και με το διορισμό της νέας Επιτροπής. Και θα ξεκινήσω με αυτά λοιπόν, που είναι σημεία που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την επόμενη εβδομάδα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα κοιτάξουν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα με την επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας. Το θετικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ε, στην Ιρλανδία και η υπογραφή της ε, Πολωνικής Προεδρίας προχώρησαν ιδιαίτερα τα πράγματα, αλλά λείπει μία χώρα. 26 στους 27 επικύρωσαν, εκκρεμεί η τσεχική υπογραφή. Στην Τσεχία εγκρίθηκε η συνθήκη από το Κοινοβούλιο, αλλά 16 γερουσιαστές ζήτησαν προσφυγή στο συνταγματικό δικαστήριο για να δουν αν είναι συμβατή η συνθήκη της Λισαβόνας με το τσεχικό σύνταγμα. Σίγουρα πρέπει να σεβαστούμε τις αποφάσεις της Τσεχίας. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει μια απάντηση, ε, μια ανοιχτή ερώτηση μάλλον, ε, στο συνταγματικό δικαστήριο και μετά από λίγες μέρες θα πρέπει να απαντήσει το συνταγματικό δικαστήριο. Ο πρόεδρος Κλάους έθεσε ορισμένους όρους για την επικύρωση και εμείς πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι όροι και τι επιφέρουν. Η συζήτηση λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξαρτηθεί από όσα θα συμβούν στην Τσεχία. Όλες οι διαδικασίες στη Τσεχία θα είναι πολύ σημαντικές για μας και για τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Όλες οι προετοιμασίες έχουν γίνει ούτως ώστε η εφαρμογή να γίνει με τον πιο διαφανή τρόπο. Θα γίνει και μία αποτίμηση της Προεδρίας για το πού βρισκόμαστε. Θα έχουμε ήδη και τις θέσεις ε, για το θέμα της Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της χρηματοδότησής της. Ε, διάβασα και την έκθεση Μπροκ σχετικά και θα εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό σήμερα το απόγευμα. Μπορώ όμως να σας πω ήδη ότι για την επόμενη εβδομάδα η έκθεση θα αποτελέσει βάση σκέψης ούτως ώστε με τη θέση σε ισχύ της ε, συνθήκης να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια επίσημη πρόταση για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσει η εξωτερική δράση και το Συμβούλιο να ξεκινήσει μια γρήγορη διαδικασία έγκρισης τους επόμενους μήνες. Τα έχουμε ήδη συζητήσει εδώ με το Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε όλη αυτή η διαδικασία συζήτησης να συνεχιστεί καρποφόρα και τις επόμενες εβδομάδε. Ένα μεγάλο θέμα που θα συζητήσει το Συμβούλιο είναι οι κλιματικές αλλαγές και για την ε, χρηματοδότηση των ε, σχετικών ε, γραμμών για την προστασία του περιβάλλοντος, ούτως ώστε να παίζει η Ευρώπη έναν αρχηγικό ρόλο στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Εχθές το ΕΚΟΦΗΝ κατέληξε σε ε, μάλλον ε, συζήτησε ορισμένες προτάσεις και αποφάσισε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά για να προχωρήσουμε. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ούτως ώστε όλη αυτή η διαδικασία να μην καθυστερήσει. Σε αυτή τη φάση γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες είναι οι δυσκολίες που μας περιμένουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει ότι άμα συμφωνήσουμε στη χρηματοδότηση θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα σε όλες τις ε, διαπραγματεύσεις. Αν όλοι συνεργαστούμε θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στην Κοπενχάγη. Τώρα, αυτή τη στιγμή συνεδριάζουν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος για να διαμορφώσουν ακριβώς τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διαπραγμάτευση. Και οι προτάσεις αυτές θα ορίσουν και μία στρατηγική για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στο στόχο μας για την μείωση των εκπομπών για το μέλλον. Τα συμπεράσματα του, του Συμβουλίου θα συμπεριλαμβάνουν και τα απορίσματα της συζήτησης για τις εκπομπές στους ε, τομεακούς μηχανισμούς, δηλαδή ναυτιλία, δάση και θα εξετάσει επίσης και το νέο πλαίσιο ενός, μηχανισμού για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Έχει προταθεί ένα σχέδιο πολύ φιλόδοξο, δημιουργία δηλαδή ενός μηχανισμού που θα περιφρουρεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα για τις τράπεζες, για τις ασφάλειες και τις μετοχές. Έχει κατατεθεί σχετικά μία νομοθετική πρόταση και αυτή είναι και μία από τις μεγάλες προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα ιδιαίτερα φιλόδοξο, διότι στα τέλη της χρονιάς θέλουμε συμφωνία για όλο αυτό το πακέτο και είμαστε πολύ ευτυχείς που το ΕΚΟΦΗΝ προχώρησε ιδιαίτερα εχθές καταλήγοντας σε μια πολιτική συμφωνία για τη δημιουργία αυτού του οργάνου περιφρούρησης, χωρίς φυσικά όμως να προδικάζονται οι συζητήσεις στα Εθνικά Κοινοβούλια. Η Προεδρία, η Σουηδική Προεδρία, ανέλαβε να συνεχίσει το διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονε, διότι θεωρούμε ότι αυτό ο διάλογο λειτουργεί ιδιαίτερα εύρυθμα. Θέλουμε να ολοκληρώνουμε με αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό για να αποφύγουμε μελλοντικέ κρίσει ούτω ώστε οι επενδυτές και οι αποταμιευτέ να ξαναβρούν την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Για την απασχόληση στην Ευρώπη είναι ένα πρόβλημα που θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εμείς τελευταία είδαμε μερικά μηνύματα ανάκαμψης αλλά δεν είμαστε ακόμη σίγουροι ότι η κατάσταση θα προχωρήσει θετικά. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μέτρα κίνητρα. Θα πρέπει λοιπόν και να αντιμετωπίσουμε την κρίση αλλά και να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τους στόχους μας για την απασχόληση όπως είχαν οριστεί πριν από την κρίση. Όλα είναι πολύ σημαντικά για την ευημερία και τη συνοχή της Ευρώπης. Εμείς ήδη αναφερθήκαμε ε, στο θέμα της exit strategy της στρατηγικής εξόδου από την κρίση. Θέλουμε μια φιλόδοξη πολιτική για την υλοποίηση των όσων συζητήθηκαν στο άτυπο Συμβούλιο του Γκέτεμπορκ, Συμβούλιο Κοφίν. Επίσης, την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσουμε το θέμα των ενεργειακών υποδομών, των διασυνδέσεων των δικτύων και της αντιμετώπισης των ενεργειακών κρίσεων. Επίσης, το Συμβούλιο θα εγκρίνει μία στρατηγική για την Βαλτική. Η συζήτηση έγινε το Σεπτέμβριο. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα εγκρίνουν τα συμπεράσματα της Προεδρίας. Αυτή η στρατηγική θέλει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που μας επιβάλλει η δημιουργία της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη και ελπίζουμε ότι θα εμπνεύσει σχέδια για άλλες μακροπεριφέρειες της Ευρώπης. Επίσης θα παρουσιάσουμε και τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας που γεννήθηκε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε να υλοποιήσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα αυτήν τη στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να προσεγγίσουμε τους στρατηγικούς μας στόχους. Επίσης θα εξετάσουμε και την πρόοδο στην υλοποίηση των συμπερασμάτων που είχαμε εγκρίνει παλιότερα για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης στην Μεσόγειο. Είχαμε το σχέδιο πιλότο για τη Μάλτα. Επίσης θα συζητηθεί το θέμα του, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ασύλου. Θα συζητηθεί και το θέμα της Τουρκίας και το ρόλο που παίζει στον χώρο αυτό. Θα συζητηθεί το θέμα της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών. για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις προσπάθειές μας για την υλοποίηση, την πλήρη υλοποίηση του Frontex. θα συζητηθεί επίσης το θέμα των εξωτερικών δράσεων στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν. τον Σεπτέμβριο είχε συζητηθεί το ζήτημα στην άτυπη συνεδρίαση. Την επόμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών η Ευρώπη θα δει πως μπορεί να συμμετέχει πιο δυναμικά στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν. Το σχέδιό μας για την περιοχή αυτή θα πρέπει να υλοποιηθεί τον νωρίτερο δυνατό. Οι στρατιωτικές λύσεις δεν είναι αηφόρες λύσεις. Για να έχουμε ασφάλεια πρέπει να έχουμε και οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει να έχουμε ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και των δημοκρατικών θεσμών. Ο ρόλος μας είναι πάρα πολύ σημαντικός σε αυτή την περιοχή. Υπάρχουν περιφερειακές προκλήσεις, αλλά πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιομορφίες της κάθε χώρας, δηλαδή και του Αφγανιστάν και του Πακιστάν. Είμαι έτοιμη να ακούσω τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. που μας παρουσιάσατε το πρόγραμμα του Συμβουλίου, ο κύριος Πρόεδρος της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Προεδρία του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Μετά από αυτά που είπε η κυρία Μάλστρομ εξ ονόματος Συμβουλίου, θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα, τη συνθήκη της Λισαβόνας και τα θεσμικά, από τη μία, και την καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών με τη διάσκεψη της Κοπεχάγης από την άλλη. Το Συμβούλιο θα πάρει την τελική απόφαση για την ε, εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο πράγμα η εφαρμογή μιας νέας συνθήκης πάντοτε, αλλά κάθε φορά που χρειάστηκε η νέα συνθήκη είχε σαν στόχο μια πιο δημοκρατική λειτουργία της Ευρώπης. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την νέα συνθήκη και για την υποστήριξη του Ιρλανδικού λαού. Η επικύρωση από την Πολωνία ολοκληρώνεται και μπορούμε τώρα να πούμε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν δημοκρατικά δεχτεί τη συνθήκη αυτή. Περιμένουμε βέβαια την Τσεχία, αλλά είναι θέμα διαδικαστικό και σεβασμού των, του δημοκρατικού χαρακτήρα τους των διαδικασιών αυτών. Ελπίζω να μην τεθούν τεχνητά εμπόδια και καθυστερήσεις στις διαδικασίες αυτές και στην Τσεχία. Έχω ήδη πει στο Κοινοβούλιο πόσο σημαντικό είναι να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και να γίνει ό,τι μπορεί να γίνει για να επιταχυνθεί η επικύρωση και εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας για να εφαρμοστούν τα αιτήματα και του Κοινοβουλίου αυτού τα οποία είχε εκφράσει και όταν ενέκρινε τον διορισμό μου ως Προέδρου της Κομισιόν για να είναι η λειτουργία της Ευρώπης πιο αποτελεσματική. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Συμβούλιο πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, να αναγνωρίσει ότι είναι επίγουσα η επικύρωση της συνθήκης, γιατί όσο δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί όπως πρέπει, θα υπάρχει μεγάλο κόστος για ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει βέβαια να είμαστε ήδη έτοιμοι για την εφαρμογή της συνθήκης, Ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί μαζί μας για να εφαρμοστεί στο δυνατόν συντομότερα η συνθήκη. Έχει ήδη αρχίσει την προετοιμασία τονίζοντας τα σημαντικότερα στοιχεία όπως την, Ευρωπαϊ... την πρωτοβουλία των πολιτών η έκθεση Μπροκ ακριβώς τονίζει αυτά τα σημεία ώστε το κοινοτικό σύστημα να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και να είναι πιο αποτελεσματικό. ξέρω ότι έχουν ακουστεί ανησυχίες ότι μήπως υπάρξει κάποιος φραγμός στη λειτουργία των θεσμών από την work closely with all institutions ναι. η εξωτερική υπηρεσία τελικά δημιουργήσει φραγμούς της λειτουργίες, αλλά δεν το πιστεύω, διότι και τα τρία όργανα είναι διατεθειμένα να συνεργαστούν έτσι ώστε οι εξωτερικές δράσεις της Ένωσης να είναι κάτι παραπάνω από το απλό άθροισμα των μερών της. η σύνδεση που έχει το Συμβούλιο με τις ε, κυβερνήσεις των κρατών είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για πιο αποτελεσματική επίτευξη των ενωσιακών στόχων. Η ε, υπηρεσία αυτή θα είναι λοιπόν ένα εργαλείο για μια πιο ενωμένη Ευρώπη. Ταυτόχρονα πρέπει να δει το Συμβούλιο τι γίνεται με την κρίση και ποια είναι οι επιπτώσεις της στην ανεργία ώστε να γίνει ό,τι μπορεί να γίνει για να εφαρμοστούν όσο το δυνατόν συντομότερα οι προτάσεις της Κομισιόν για τη ε, ναι, επιτήρηση και παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών θεμάτων. Το άλλο σημαντικό θέμα βέβαια είναι η Κοπεχάγη. Η επιτυχία της διάσκεψης αυτής ενδιαφέρει πολλούς Ευρωπαίους και θα αποτελέσει δοκιμή για όλους. Η πρόοδος των διαπραγματεύσεων παραμένει βέβαια αργή. Δεν πρέπει όμως να χαθεί η ορμή, η αρχική ορμή, της, ορμή τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι για να αντιμετωπίσουμε σφαιρικά τα πράγματα χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα. Συγκεκριμένες ιδέες και για χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Μέχρι το 2020 υπολογίσαμε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα χρειαστούν 100 παραπάνω δισεκατομμύρια το χρόνο. Οι αναδυόμενες οικονομίες ιδιαίτερα θα μπορέσουν να καλύψουν μεγάλο τμήμα της ανάγκης αυτής, αλλά χρειάζεται πρόσθετη χρηματοδότηση και από την Ένωση. Στο πρόγραμμα της Κοπεχάγης δεν αναφέρονται μόνο κλιματολογικές αλλαγές που είναι βέβαια το κυριότερο θέμα, αλλά και θέματα αναπτυξιακά. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και πρέπει εδώ η Ευρώπη να αναλάβει δεσμεύσεις όλοι γνωρίζουμε ότι όσο περισσότερο περιμένουμε τόσο υψηλότερο θα είναι το κόστος. Και εδώ το Συμβούλιο πρέπει να βρει ευρηματικές λύσεις και ενωτόμες λύσεις ώστε να υπάρξει μια ενωμένη Ευρώπη για την καταπολέμηση των επιπτώσεων των κλιματολογικών αλλαγών. Να δείξει η Κοπεχάγη δηλαδή ότι έχει αρχίσει ήδη να εφαρμόζεται η μείωση των εκπομπών. Αυτό θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να φανεί ότι η συνθήκη της Λισαβόνας αρχίζει ήδη να λειτουργεί και επιφέρει συγκεκριμένα ωφέλη στους πολίτες. Και έτσι επανέρχομαι, χρειάζεται γι' αυτό ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο. Η συνθήκη της Λισαβόνας είναι η πρώτη ευρωπαϊκή συνθήκη μετά τη μεγάλη διεύρυνση. Η πρώτη συνθήκη είχε συγγραφεί σε μια διαιρεμένη Ευρώπη. Πρέπει όμως τώρα οι θεσμοί της διευρυμένης Ευρώπης να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την καινούργια αυτή πραγματικότητα με τη συνθήκη ακριβώς της Λισαβόνας για να υπάρξουν πιο αποτελεσματικά ωφέλη για τους πολίτες στην Ευρώπη των 27. Γι' αυτό βέβαια χρειάζεται και πολιτική θέληση και ελπίζω ότι στο τέλος του μηνός το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επιδείξει αυτή την πολιτική θέληση στην Κοπεχάγη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε της Εκτελεστικής Επιτροπής, για τις πολιτικές ομάδες θα δώσουμε το λόγο καταρχήν στον κύριο Ντόλ, Πρόεδρο της ομάδας του ΕΛΚΟΜ. Κυρία κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ομάδα του ΕΛΚΑ από το επόμενο διάσκεψη κορυφής περιμένει να τελειώσει η μακρά περίοδος αβεβαιότητας για τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης και να δώσει την απαραίτητη όρμη για τον διορισμό της Νέας εκπαιδευτική Επιτροπής αλλά και μια σταθερή Προεδρία του ε, Συμβουλίου και τον είπα το εκπρόσωπο προβλέπει συνδείξη Λισαβόνα θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ναι. αναλάβει τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσει να ξαναδώσει μια οικονομική όθηση και να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει θέσει απασχόληση. Γιατί η κρίση δεν θα έχει τελειώσει εφόσον δεν θα έχει επανέρθει η κοινωνική ισορροπία. Για τα θεσμικά όργανα, θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι με την απόφαση του Πολωνού Προέδρου να υπογράψει τη συνθήκη, έχουμε όλε τι χώρε εκτό από μία που άνοιξαν το δρόμο για να μπορέσει επιτέλους να προχωρήσει η Ευρώπη. Στις 27 Οκτωβρίου, δύο μέρες πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ε, το Συντασματικό Δικαστήριο της Τσεχίας θα μελετήσει το κατά πόσον η συνθήκη αυτή είναι συμβατή με το Σύνταγμα της εν λόγω χώρας. Βέβαια θα σεβαστούμε την απόφαση αυτή, όποια και αν είναι. Απ' την άλλη μεριά, η ομάδα μου λυπάται που ο Τσέχος Πρόεδρος, ενώ η ε, το κοινοβούλιο του ε, υπερψήφισε τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας έχει μία πρόφαση τώρα για να μην υπογράψει. Ίσως να του δώσουμε κάποιες διαβεβαιώσεις για κάποια σημεία της συνθήκης, αλλά δεν πρέπει να ξαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Χαιρετίζω την απόφαση αυτή η ομάδα του ΑΛΚ περιμένει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην δεχθεί αυτά, αυτούς τους ελιγμούς. Όλοι οι λαοί έχουν προσυπογράψει τη συνθήκη και θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Εφόσον η συζήτηση στην Ευρώπη ε, κα, ε, στη συζήτηση στην Ευρώπη επικρατεί η θεσμική συζήτηση, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά, ούτε κοινωνικά, ούτε οικολογικά τα θέματα αυτά δεν θα εξεταστούν με την απαραίτητη σοβαρότητα και ταχύτητα. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ε, <clears throat> δεν προχωράμε. Κάνουμε σημειωτό βήμα. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εκφραστεί κατά το δυνατόν πριν από τα τέλη του έτους πάνω στις ε, θέσεις που θα χορηγηθούν στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο. Επίσης, η ομάδα του ΕΛΚ περιμένει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συγκεκριμένου προσανατολισμού για την οικονομική πολιτική ακολουθώντας και τις αποφάσεις του Πιτσμπουργκ που έδωσε κάποια αμφίβολα αποτελέσματα και βλέπουμε στον τύπο ότι συνεχίζεται η κατάσταση να μην έχει γίνει τίποτα. Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς δραστηριότητες για να υπάρχουν επενδύσεις και στην έρευνα. Η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει ό,τι χρειάζεται για να υπάρχει ε, ισότιμο εμπορικό περιβάλλον και επίσης περιμένω μια προσαρμοσμένη πολιτική για το κλίμα που βρισκόμαστε σε δύο μήνες από την Κοπεχάγη. Και αναρωτιέμαι ποια θα είναι η πίεση που μπορούμε να ασκήσουμε στη ΣΥΠΑ, στην Κίνα και σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μια ευγενική και μετριασμένη πίεση ή μια μέγιστη πίεση. Χαίρομαι που είναι ηγέτης η Ευρώπη στο θέμα αυτά, αλλά δεν μπορεί να είναι η μόνη που θα καταβάλει προσπάθειες για να καταπολεμήσει την υπερθέρμανση του πλανήτη. 50 μέρες μένουν για την Κοπενχάγη. Δεν είναι πολλέ ίσως, αλλά αρκούν αν θέλουμε να προχωρήσουμε σωστά και με βοστικότητα. Και ελπίζω, κύριε Πρόεδρε του Κομισιόν, να, κύριε Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, να μας πείτε πώς θα εκμεταλλευτείτε τις 50 αυτές μέρες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου θα είναι μια στιγμή κλειδί για την Ευρώπη, για τις ε, δεσμεύσεις που αναλάβει, για την οικονομία, για τα κοινωνικά θέματα και να ξεπερέσει τις θεσμικές διαμάχες. Η ομάδα μου κάνει έκκληση να αναλάβει κάθε ένα από τα 27 κράτη-μέλη τις ευθύνες του. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα Εξ ονόματο τη Σοσιαλιστική Ομάδα, ο κύριο Χάνε Φόβοντα έχει το λόγο. Äh, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε τη Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, πριν αναφερθώ συγκεκριμένα στο θέμα αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ στα σύντομα στην Κοπεχάγη. Έχετε δίκιο, κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριο Πρόεδρο τη Επιτροπή, το τόνισε. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικέ αποφάσει που πρέπει να πάρουμε προ την κατεύθυνση τη Κοπεχάγη και χρειαζόμαστε θεσμευτικού ε, στόχους, όχι γενικές δηλώσεις. Δεν αρκεί αυτό, μια που οι Αμερικανοί δεν έχουν προχωρέσει με την ε, νομοθετική τους διαδικασία και πολλά θα πρέπει να γίνουν και μετά την Κοπεχάγη, αλλά για το τέλη της ε, διαδικασίας θα πρέπει να υπάρχουν δεσμευτικοί όροι. Τώρα, όσον αφορά τις ε, αγορές και την οικονομική κατάσταση. Είναι πραγματικά προκλητικό και εξωφρενικό όλες αυτές οι οι προμοδοτήσεις που δίνονται στους ανθρώπους σε αυτό το τομέα. Στη ΣΥΠΑ ιδίω. Κανένα δεν καταλαβαίνει όμω γιατί γίνεται αυτό όσον αφορά και την ευθύνη που πρέπει να αναλάβουν οι άνθρωποι αυτοί έναντι των πολιτών. Έχετε δίκιο, κυρία Πρόεδρε, από του Συμφουλίου, ότι κυρίω το θέμα τη απασχόληση θα πρέπει να μα απασχολήσει. Δεν είναι το θέμα το να μην σταματήσουμε και να μην τερματίσουμε τις, ε, τα κίνητρα που δίνουμε αυτή τη στιγμή. Όχι, πρέπει να δώσουμε νέα κίνητρα, να αποφασίσουμε νέα στοιχεία για να προωθήσουμε την απασχόληση. Ο πρόεδρος της ε, Κομισιόν αναφέρθηκε χθε πολύ προσεκτικά σε αυτό και χαίρομαι που φαίνεται ότι διαφαίνεται αυτή τη στιγμή μία συνενετική πολιτική για το θέμα της απασχόλησης. Δύο λόγια για τη Λισαβόνα. Καταρχήν για την ε, απουσία της υπογραφής του Βακλαφ Κλάους ελπίζω θα υπάρχει μια θετική απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου. Μου φαίνεται απαράδεκτο να χρησιμοποιούν τώρα οι αποφάσεις μπενές για να υπάρχει καθυστέρηση αυτή της υπογραφής. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους από τη Δημοκρατία Θυμάστε, τότε είσαστε μεταξύ μας κύριε Προεδρεύουσα, είχαμε αναθέσει μία έρευνα για τα διατάγματα αυτά Μπένεσ. Πλειοψηφικά αποφασίσαμε ότι αυτά τα διατάγματα δεν είναι ε, εμπόδιο, δεν μπορούν να είναι εμπόδιο για την ένταξη της ηχείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν είπαμε ότι δεν παρεμποδίζουν την έναρξη της Ευρωπα... της... στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Αιχικής Δημοκρατίας, δεν μπορούν τώρα τα ίδια διατάγματα μπαίνες να χρησιμοποιηθούν για να μην δοθεί η υπογραφή αυτή. Θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Η συνδίκη της Λισαβόνας έχει κυρίως δύο στόχους. Περισσότερη δημοκρατία στην Ευρώπη, περισσότερη και κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν θέλετε γιατί δεν είστε υπέρ της περισσότερης δημοκρατίας, δεν ναι, ξέρω. Και δεύτερον, περισσότερη αποτελεσματικότητα. Και νομίζω, κύριε Πρόεδρε ε, τη Εκτελεστικής Επιτροπής, αυτό είναι ένα σημαντικό έργο που αναλαμβάνεται για τι επόμενε εβδομάδε. Να φροντίσετε τα θέματα τα θεσμικά και τα προσωπικά να μην υπάρχουν εμπόδιο. Ο κύριος Μπαρόζο είπε χθε δικαίω ότι χρειαζόμαστε έναν πρόεδρο του Συμβουλίου, για τον οποίο δεν έχουμε καμία επίδραση, έναν πρόεδρο του Συμβουλίου, ο οποίος θα συνεργάζεται με την Κομισιόν και με το Κοινοβούλιο και θα εφαρμόζει την κοινοτική μέθοδο σαν επίκεντρο της διαδικασίας απόφασης του. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν χρειαζόμαστε έναν πρόεδρο του Συμβουλίου που να στολίζεται σαν παγόνι και να βγάζει κάποιους κυριακάτικους λόγους εδώ. Δεν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε κάποιον που να εργάζεται σκληρά και χρειαζόμαστε και μια εξωτερική υπηρεσία η οποία όχι μόνο θα υιοθετεί αποτελεσματικές μεθόδους κοινοτικές, αλλά που θα αναφέρεται και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δεν επιτρέπεται. Από τη δίκηση της Λισαβόνας που έχει σαν στόχο περισσότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο, να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να οδηγεί σε λιγότερο ε, κοινοβουλευτικό ε, ε, έλεγχο και να εωρείται η εξωτερική υπηρεσία αυτή υπεράνω ημών. <coughs> Και ακριβώς με τον συνάδελφο Μπρόκο συζητητή και με τον πρόεδρο της ε, Εκτελεστικής Επιτροπής συμφωνούμε απόλυτα για το θέμα αυτό. Και τονίζω ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος θα πρέπει να υπάρχει και για την εξωτερική υπηρεσία μέσω του είπα του αυτού εκπρόσωπου βέβαια και υπό τον έλεγχο του Συμβουλίου πάντα. Άρα ο Στέος Συνάλφος ξέρω ότι προσπίζεται τις ιδέες σας αυτές και ότι θα εφαρμοστεί έτσι η συνθήκη της Λισαβόνας. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερο δημοκρατικό έλεγχο και περισσότερα αποτελεσματικότητα στην εξωτερική πολιτική. Ευχαριστώ of blue card question if you want to take it. Yes, okay. Υπάρχει εδώ Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σβόμποντα καταρχήν ο κύριος Βάρντς. Tisztelt Svoboda úr, ön azt említette, hogy Κύριε Σβόμποντα, εσείς είπατε λέει ο κύριος Μπάλσο με μπλε κάρτα ότι το διάταγμα Μπένες δεν αποτέλεσε εμπόδιο, αλλά ξέρετε όμως ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις του διατάγματος Μπένες, οι οποίες ισχύουν. Όντας η Ευρώπη ένα κράτος δικαίου πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και στους Σουδίτες και στους Γερμανούς. Ναι, Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί Σουδίτες που ζουν στην Αυστρία και θα πρέπει να γνωρίσουμε τα αισθήματά τους, αλλά θα πρέπει να ξεχάσουμε το παρελθόν, να ταινίσουμε προς το μέλλον. Και το μέλλον δεν είναι τα διατάγματα του Μπένος, είναι μια ελεύθερη Ευρώπη, με ελεύθερους πολίτες που έχουν δικαιώματα που απορρέουν από, τη χάρτα βασικών δικαιωμάτων. Thank you, σας ευχαριστούμε και τώρα θα ακούσουμε εξ ονόματος της ομάδας του τον κύριο Φερχόφσταντ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Έχουν πάει τόσο μακριά ήδη τα πράγματα αλλά το τρένο φαντάζομαι ότι δεν μπορεί πια να σταματήσει. Αυτό είπε ο κύριος Κλάους και είναι η μόνη δήλωσή του με την οποία συμφωνώ ότι το τρένο έχει ήδη πάει τόσο μακριά και τόσο γρήγορα ώστε δεν μπορεί πια να σταματήσει. Πολύ σημαντική δήλωση διότι ο πρόεδρος Κλάους φαίνεται ότι δέχεται έτσι ότι δεν μπορεί τίποτε να καθυστερήσει πια την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας είναι φυσικό αν 27 κράτη την έχουν εγκρίνει και επικυρώσει να την επικυρώσει και εκείνο. Η αλλαγή αυτή στη στάση του δεν μπορεί να εξηγηθεί παρά μόνο από την κατανόηση του γεγονότος ότι όλοι είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν στην εφαρμογή της συνθήκης. Και στις επόμενες μέρες και εβδομάδες θα ελπίζω να φανεί Δηλαδή ότι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσει κανείς την επικύρωση της συνθήκης είναι, κυρία Μάλστρομ, να αρχίσει ήδη κανείς την εφαρμογή, την προετοιμασία της. Αυτό δεν είπε και εκείνος, ότι το τρένο έχει προχωρήσει. Δεν μπορεί να σταματήσει το τρένο, θα συνεχίσει το τρένο. Και γι' αυτό είναι απολύτως απαραίτητο το Συμβούλιο να επιταχύνει τις διαδικασίες να εγκρίνει το θέμα των διορισμού ας πούμε του είπα του αρμοστή αφού το τρένο είπαμε τρέχει και ο κύριος Κλάους δεν θα μπορέσει πάνω να προσυπογράψει και αν προχωρήσετε θα το κάνει και εκείνος Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, Εξωτερικής Δράσης. Ελπίζω το Συμβούλιο να καταλήξει και από αυτό όχι όμως να συμφωνήσει οτιδήποτε, να μην υπάρξει επικάλυψη γιατί υπάρχει ο φόβος ότι θα δημιουργηθούν δύο παράλληλες δομές μία από την Κομισιόν και αυτή θα αντιπροσωπεύει, αντιπροσωπεύει ήδη περίπου 6.000 υπαλλήλους και από την άλλη μια νέα υπηρεσία εξωτερικής δράσης με χιλιάδες πάλι υπαλλήλου που θα εξυπηρετούν τον ύπατο αρμοστή. Νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει μία και μόνη δομή που να ασχολείται με τις εξωτερικές υποθέσεις και όχι αυτές οι δύο παράλληλες των αντιπροσωπιών της Κομισιόν από τη μία και της εξωτερικής υπηρεσίας από την άλλη, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Πρέπει το Συμβούλιο να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά συμφωνία όπου να αποσαφηνίζεται ότι δεν θα υπάρχει επικάλυψη στις δομές αυτές και στις δραστηριότητες αυτές από τη μία με τις ε, Κομισιόν και από την άλλη με την Υπηρεσία Εξωτερικών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, εξ ονόματος των Πρασίνων, η κυρία Ρεβέκα Χάρμς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξότιμη εκπρόσωπο του Συμβουλίου και της Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την Τσεχία, καταρχήν. Μου φαίνεται πραγματικά μια ιδιαίτερη πολιτική αυθάδια πώς δρά ο κύριος Κλάος ως εκείνος που έχει χάσει το παιχνίδι Και αυτός ο άνθρωπος που δεν σέβεται καν την το τσεχικό σύνταγμα γιατί δεν σέβεται την πλειοψηφία στη Βουλή τη δική του που ενέκρινε την ε, συνθήκη της Λισαβόνα, αυτό τον άνθρωπο δεν θα πρέπει να τον ε, υποστηρίξετε όταν ζητήσει opt-out για την Τσεχία όσον αφορά την Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτός είναι ένας έχος troublemaker θα μπορούσα να πω. Ένας άνθρωπος που σπέρνει ζυζάνια. Και πραγματικά αξίζουν πολύ καλύτερα οι πολίτες της Τσεχίας. Αυτά για τον πρόεδρο Κλάους. Για το κλίμα, κύριε πρόεδρε Παρόσο. Σπάνια με βρίσκεται τόσο σύμφωνη με αυτά που λέτε όσο σήμερα. Ενθουσιάστηκα που είπατε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν την υποχρέωση με ένα ξεκάθαρο ποσό να συμβάλλουν σε αυτό το Διεθνές Ταμείο για τα αναπτυσσόμενες χώρες για την προστασία του περιβάλλοντος. Δράπηκα χθε που διάβασα ότι ο Γερμανός υφυπουργό Οικονομικών που ήταν στην, ε, στο Λουξεμβούργο είπε ήταν σαν ένα παιχνίδι πόκα. Και όταν είπε ότι στην περίπτωση αυτή δεν λέμε τι σκεφτόμαστε. Αλλά δεν πρόκειται για πόκα εδώ στην προετοιμασία της Κοπενχάγης, πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η κυρία Μέρκετ και άλλοι σημαντικοί πολιτικοί όπως έχουν πει οι πολιτικοί αυτοί, πρόκειται για τη σημαντικότερη πρόκληση που έχουμε όλοι εμείς που ζούμε σε αυτή την γη. Εκατό δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να είναι διαθέσιμα μετά το 2020 για να βοηθηθούν τα αναπτυσσόμενα κράτη να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που θα αναλάβουν για την προστασία της κλιματολογικής. Για μια χώρα σαν τη Γερμανία θα πρόκειται για μετά το 2020 3 δισεκατομμύρια σε σχέση με αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή στο, για την προστασία του χρηματοπιστωτικού τομέα δεν είναι τίποτα τα χρήματα αυτά και πραγματικά ντρέπομαι που ε, διακυβεύουν την αποτυχία στην Κοπενχάγη με τα παιχνίδια αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως διαπραγματεύτηκε χθε στο Λουξεμβούργο δεν είναι η ατμομηχανή, δεν είναι ο ηγέτης στην προστασία διεθνώς του κλίματος αλλά είναι εκείνη που παρεμποδίζει τα πράγματα και παρακολουθούν από όλο τον κόσμο το τι γίνεται στο Λουξεμβούργο σήμερα, τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Σας παρακαλώ κύριε Μπαρόζο, παραμείνετε σε αυτή τη γραμμή της Κομισιόν. Η γραμματοδότηση θα πρέπει να προετοιμαστεί τώρα διαφανώς. Εδώ και δύο χρόνια από τον Πάλι ήδη εξετάζεται το θέμα και θεωρώ κύριε Μάρστρομ ότι οι Σουηδοί πολύ καλά διαπραγματεύονται και σας παρακαλώ να σεβαστείτε και την ψήφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί πρόκειται για δύο μειώσεις ε, για το διοξείδιο του άνθρακα κατά 30%. Εάν δεν έχουμε τη χρηματοδότηση αυτή δεν θα το πετύχουμε ποτέ. Μία τελευταία πρόταση. Έχω προβλήματα με την αξιοπιστία της ε, Σουηδικής Προεδρίας. Θα πρέπει η κρατική εταιρεία Vattenfall να φροντίσετε να μην χρησιμοποιεί σε όλη την Ευρώπη άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η στρατηγική της κρατικής επιχείρησης Βάτεφαλ έχει σε αντίθεση με την καλή σας φήμη στα κλιματολογικά θέματα. και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η προσφυγή που έκανε η Βάτα κατά της κυβέρνησης της Γερμανίας που ήθελε να της επιβάλλει κάποιες περιβαντολογικές ε, ε, διατάξεις σας παρακαλώ να αποσυρθεί έχετε εκεί ένα πρόβλημα και φροντίστε να απειληθεί πριν πάτε στην Κοπεχάγη Πρόεδρος Διακόπτη σας ευχαριστώ πάρα πολύ Παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο σας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίση, κάποιος άλλος με μια μπλε κάρτα έχει ζητήσει να μιλήσει. Δεν θα δώσω σε καθέναν τη δυνατότητα να μιλήσει. Θα υπάρχει λοιπόν και άλλη μια πρόταση ίσως. Ε, Επόμενος μιλητή λοιπόν, ο κύριο Τιμόθεος Κίρκοπ. Πρόεδρε, Καταρχήν συγχαίρω τη Σουηδική κυβέρνηση για την προεδρία της γενικότερα, ιδιαίτερα όμως για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται αυτά τα σημαντικά θέματα των κλιματολογικών αλλαγών και της χρηματοπιστωτικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Χρειάστηκε η Προεδρία να αντιμετωπίσει και το θεσμικό πρόβλημα, κυρίως τη συνθήκη της Λισαβόνας. Βέβαια τα θεσμικά δεν είναι προτεραιότητα των πολιτών. Το πρόγραμμα της Λισαβόνας τους ενδιαφέρει, όχι η συνθήκη τόσο πολύ. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης με πρωτεύοντα διεθνή ρόλο. Και αυτά μέχρι το 2010. Αν είχε επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα έβλεπε ο κόσμος ότι γίνεται κάτι απτό. Και όμως μέχρι τώρα το πρόγραμμα της Λισαβόνας αποτελεί αποτυχία. Γιατί δεν είμαστε σε θέση να έχουμε αποτελέσματα απτά για τους πολίτες. Γιατί ακούμε τόσα θετικά που δεν εφαρμόζονται όμως. Τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά κύριε Πρόεδρε είναι όλα αυτά. Πρέπει να γίνονται όλα αντιληπτά και από τους απλούς ανθρώπους. Η δημιουργία των θέσεων εργασίας δεν πρέπει να είναι εργασίας πρωθυπουργών και προέδρων συμβουλίου ή διαφόρων αφιθιονάδος των διεθνών ταξιδιών. Αυτά τέτοιου είδους θέσεις δεν βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε καμία χώρα ούτε λύνουν το πρόβλημα της κρίσης που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες. Οι θεσμικές αλλαγές δεν βοηθούν την αντιμετώπιση των κλιματολογικών τιούτων και γι' αυτό οι μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης πρέπει να λυθούν με πρακτικό και απτό τρόπο. Χιλιάδες σελίδες κειμένων γράφονται που δεν μπορεί να τις καταλάβει ο πολίτης γιατί είναι δυσνόητες και έτσι απλώς καταναλώνονται δέντρα τα οποία πρέπει να προστατεύσουμε μάλιστα. Πώς θα σώσουμε τις επόμενες γενναίες. Δεν συμμερίζονται όλοι τον ενθουσιασμό άλλων για του, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. όλα αυτά κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ελπίζω ότι η Σουηδική Προεδρία θα κατορθώσει στον υπόλοιπο χρόνο της να δείξει σε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και πολίτες ποια είναι τα κυριότερα θέματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Δηλαδή, την οικονομία της Ευρώπης και την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Τους εύχομαι καλή επιτυχία και ευχαριστώ για το μέχρι τώρα έργο τους. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα, επόμενος ομιλητής, εξ ονόματος της ομάδας της ΓΚΟΕ, θα είναι ο κύριος Λοθάριος Μπίσκι. Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε από το Συμβουλίο, κύριε Πρόεδρε της Εκθεστικής Επιτροπής, εδώ και τρεις μήνες συζητιέται το θέμα του ατόμων, το θέμα ε, που θα διοριστούν ε, το θέμα της συνθήκης της Ρισαβόνας. Θέλουμε καταρχήν την πρόθεση της κοινωνικής Ευρώπης. Θέλουμε αφοπλισμό και τρίτον περισσότερη άμεση δημοκρατία και όχι μια ελίτ Ευρώπη θα πρέπει να υπά... Ε, ασχοληθούμε με την ουσία. Ενώ συζητάμε για ονομασίες και θέσεις, πολλοί παραμένουν άνεργοι. Σώζονται οι τράπεζες βέβαια. Ταυτόχρονα ο πρόεδρος κ. Παρόζο ζητά σύντομα να εγκαταλείψουμε το πρόγραμμα ε, το συγκυριακό το 2011 και των σχετικών ε, προγραμμάτων κρατομενών. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθούν οι μισθοί, θα σημειωθούν οι συντάξεις, θα μειωθεί η κοινωνική προστασία, θα αυξηθούν οι φόροι καταναλωτικοί, δεν θα υπάρχουν πια συλλογικέ συμβάσει, Παράδειγμα, παράδειγμα από τη Γερμανία. Υπάρχει απεργία αυτή τη στιγμή στη Γερμανία όσον αφορά τον κλάδο καθαρισμού κτηρίων. Αυτά είναι τα τα προβλήματα που θα πρέπει να απασχολήσουν το Συμβούλιο. Ανταυτού συζητιώνται συμπληρωματικέ ρήτρε για τις συνθήκη τη Αβώνα που θα μπορέσουν να κινήσουν τον Τσέχο πρόεδρο για να υπογράψει. Αν τα πράγματα είναι τόσο απλά, εντάξει, Αγαπητή αρχή και κρατών και κυβερνήσεων, κάθε το. Αλλά για σκεφτείτε και για μια κοινωνική ρήτρα πρόοδου στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Θα ήταν καλό και αυτό. Στην αρχή της ε, θητείας υπήρχαν πολλές καλές προτάσεις για μια πιο κοινωνική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ αυτών ένα νέο πρόγραμμα ε, συγκυρίας για την Ευρώπη και αηφόρο οικολογική ανάπτυξη. Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Απασχόληση ζητήθη ισότιμια των μισθών, καλύτερη όρια εργασίας, αυξημένη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Η αηφορία των κοινωνικών και συνταξιακών συστημάτων θα έπρεπε επίση να εξασφαλιστεί. Προ το παρόν, ούτε στην πολιτική των κρατών μελών, ούτε στην πολιτική της Κομισιόν, βλέπω κάποια στρατηγική προ την κατεύθυνση αυτών των στόχων. Βέβαια το Συμβούλιο θα πρέπει να εξετάσει τους διορισμούς των νέων επιτρόπων και τις ενδεχόμενες αλλαγές ε, βάσει τη συνθήκη της Αβώνας. Αλλά θα πρέπει να εξεταστούν τα εν λόγω προβλήματα που ανέφερα και η εφαρμογή τους. Η δική μου ομάδα θα εξαρτήσει την ψήφο της για τους επιτρόπους από την πρόοδο στα θέματα αυτά. Ε, ε, Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φάλατ για την Ευρώπη της Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Είπατε το πρωί κύριε Πρόεδρε ότι όλα τα κράτη έχουν δημοκρατικά εγκρίνει και επικυρώσει τη συνθήκη. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Και στη Βρετανία δεν έχει γίνει δημοψήφισμα και μέχρι να γίνει εγώ δεν αρνούμε ότι επικυρώθηκε δημοκρατικά. Ο πρόεδρος Κλάους δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνει την επόμενη εβδομάδα. Ξέρω ότι όλοι τον μισείτε διότι πιστεύει στην εθνική δημοκρατία. Τι κάνει όμως, απλώς υπερασπίζεται τα ε, τσεχικά εθνικά συμφέροντα. Φοβάται τα γερμανικά συμφέροντα επί των Σουδητών και έχει απολύτως δίκιο να το φοβάται. Να επιμένεις πρόεδρε Κλάους και άμα δεν σου δώσουν αυτό που θέλεις μην υπογράφεις. και να ξαναγίνει δημοψήφισμα σε 25 πλέον χώρες μέλη. Μόνο αυτό θα ήταν δημοκρατική διαδικασία. Φαντάζομαι ότι πόσο θέλετε να γίνει δημοψήφισμα στη Βρετανία. Αναρωτιέμαι, στο τέλος της Συνόδου, τι θα δημιουργηθεί ένας Ευρωπαίος αυτοκράτορ και ποιος θα είναι, ο Τόνι Μπλερ. Εγώ καταλήγω ότι Θέλω τον Τόνι Μπλερ να τον οδιορίσετε. Είναι εκείνο που κατήργησε τη Βρετανική επιστροφή των 2 δισεκατομμυρίων και δεν την αντικατέστησε με τίποτε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φανερό ότι το βραβείο για εθνική μειοδοσία και προδοσία είναι πολύ υψηλό. Να διορίσετε τον Τόνι Μπλερ για να φανεί από το λαό ότι δεν μετρούν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι αλλά οι προδότες της εθνικής δημοκρατίας ότι αυτοί παίρνουν τις υψηλότερες θέσεις δώστε μας τον Τόνι Μπλερ σας παρακαλώ ως πρώτο πρόεδρο της Ευρώπης ευχαριστούμε πολύ και τώρα ο κύριος Ντότζ η κυρία Ντότζ δεν ήταν αναπάντεχο, αν και είναι απογοητευτικό, ότι όλοι επιμένουν για την ταχύτερη δυνατή εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας. Ξέρω ότι δεν συμφωνείτε όλοι, αλλά εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει, έπρεπε να γίνει δημοψήφισμα για τη συνθήκη. Και δεν καταλαβαίνω γιατί και οι συντηρητικοί και οι εργατικοί δεν το έκαναν. Σήμερα όμως θα ήθελα, κυρία Υπουργέ, να τονίσω ιδιαίτερα το θέμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης που συνεχίζει να μας πλήττει. Εχθές το βράδυ ο κύριος Μέρτον Κίνγκ που διευθύνει την τράπεζα της Αγγλίας είπε ότι οι δανειοδοτήσεις του κράτους προς τις τράπεζες πλησίαζε το 1 τρισεκατομμύριο λίρες. Είπε μάλιστα ότι ποτέ δεν είχαν δοθεί τόσα πολλά χρήματα από τόσο λίγους σε τόσο λίγους. Αυτό είναι η μόνη μεταρρύθμιση που έχουμε δει. Και είπε ότι υπάρχει ένα ηθικό δίλημα στην καρδιά της κρίσης αυτής. Δηλαδή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα γνώριζαν ότι είχαν υπερβολική σημασία για να τα αγνοήσουν και ότι οι φορολογούμενοι και στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού θα χρειαζόταν πάντοτε να πληρώσουν την ύφη, όποια και να ήταν η κρίση. Αυτή είναι πολύ σοβαρή κατηγορία και προέρχεται από εκπρόσωπο των τραπεζικών, του τραπεζικού κόσμου. Πρέπει το ηθικό αυτό δίλημα να λυθεί κάπως. Κυρία μου σας παρακαλώ ξεπεράσατε το χρόνο σας. Θα με συγχωρείτε κυρία μου αλλά ξεπεράσατε είπα το χρόνο σας. Μην ξεπερνάτε παρακαλώ συνάδελφοι γιατί θα διακόπτω. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο του Συμβουλίου, την κυρία Μάλστρομ. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να τοποθετηθώ και φυσικά θα παραμείνω σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Κύριε Φερχόφστατ, εγώ πιστεύω ότι θα έρθει κάποια στιγμή η κατάλληλη στιγμή. Η Σουηδική Προεδρία έχει ιδιαίτερα στενές επαφές με την Τσεχική ε, κυβέρνηση και ελπίζουμε ότι θα σας δώσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα τις καλές πληροφορίες και τα καλά νέα. Για τους ε, διορισμούς ε, περιμένουμε να γίνουν οι διορισμοί, θα φτιάξουμε έναν κατάλογο πλήρη και ο οποίος θα σας δοθεί το συντομότερο δυνατόν. Για τη διάσκεψη κορυφής θα ληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες αποφάσεις ε, μπορούν να ληφθούν και όταν θα έχουμε όλες τις επικυρώσεις θα θέσουμε σε ισχύ τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους ε, τους βουλευτές ε, για την υποστήριξη που δώσανε σε έναν από τους βασικούς στόχους της Σουηδικής Προεδρίας ναι, η επιτυχία της διάσκεψης ε, της ε, Κοπενχάγης. Είναι μια τεράστια πρόκληση για την Ευρώπη. Υπάρχουν ε, και οικονομικά προβλήματα. Πρέπει να αναλάβουμε εμείς τις οικονομικές μας ευθύνες για να στείλουμε ένα παγκόσμιο μήνυμα. Έχουμε επαφές και με άλλους βασικούς πρωταγωνιστές όλη την ιστορία, τους Ρώσους και τους Αμερικάνους με τους οποίους έχουμε ραντεβού στην Κοπεχάγη για διμερείς επαφές. Έχουμε τη συνεδρίαση της Βαρκελόνης σε 10 μέρες. Έχουμε λοιπόν πολλές ευκαιρίες για τη συζήτηση. Εγώ δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι τώρα, αλλά ελπίζω, όντας αισιόδοξη, ότι θα καταφέρουμε κάτι πριν από την Κοπεχάγη, γιατί το προσδοκούν οι, πάλι, οι πολίτες όλου του κόσμου. Ελπίζουμε επίσης ότι θα έχουμε αποτελέσματα για τη διαχείριση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Υπάρχει αυτό το σχέδιο για τη δημιουργία του οργανισμού παρακολούθησης το συντομότερο δυνατό για να μπορεί να κρούει τον συναγερμό και να διαχειρίζεται τις κρίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα κερδίσει ποτέ την εμπιστοσύνη των πολιτών της αν δεν λύνει τα προβλήματα που τους απασχολούν. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν λύσεις στη διάρκεια όλων αυτών των συζητήσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ. Τώρα ο κύριος Μπαρόσο. Νομίζω ότι ο πρόεδρος του Ελκο, ο κύριος Δόλ και η κυρία Άρμς έθεσαν μερικά πολύ σημαντικά ζητήματα. Πώς μπορούμε εμείς να έχουμε επιτυχίες στην Κοπενχάγη, κυρίως όταν έχουμε άλλους εταίρους που δεν καταβάλουν τις ίδιες προσπάθειες. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες, διότι υπάρχει μία έλλειψη φιλοδοξιών από ορισμένες αναπτυγμένες χώρες ε, ως προς την ανάληψη δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών Υπάρχουν αντιστάσεις από τις μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να μπουν μέσα, στα μέσα στο γενικό πακέτο και τα εθνικά του σχέδια για τη μείωση και επίσης δεν υπάρχουν αξιόπιστες οικονομικές απαντήσεις. Τι να κάνουμε... Δεν είναι ώρα για την Ευρώπη να μειώσει τις φιλοδοξίες της, διότι έτσι θα δώσουμε προσχήματα σε όλες τις ε, αρνητικά διακείμενες ε, δυνάμεις για να μην, καταλάβουν, να μην καταβάλουν προσπάθειες. Εμείς πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε τον ηγετικό μας ρόλο. Και απαντώ εδώ στον Σοζεφ Ντόλ, η οικονομική μας βοήθεια είναι επιλεκτική και υποθετική. Εμείς θα βοηθήσουμε αυτούς που θα καταβάλουν προσπάθειες. Το να μειώσουμε τις φιλοδοξίες μας θα ήταν λάθος. Θεωρώ ότι υπάρχουν πιθανότητες επιτυχίες της Κοπενχάγης. Υπάρχει και ένα θετικό μήνυμα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε μπήκαν στην, ε, στη διαπραγμάτευση πριν από μερικά χρόνια. Απουσίαζαν οι Αμερικάνοι. Η Αυστραλία εξήγηλε φιλόδοξους στόχους, όχι δεσμευτικούς αλλά φιλόδοξους. Η Κίνα, το Μεξικό, η Βραζιλία, η Νότια Κορέα εξήγηλαν φιλόδοξα εθνικά σχέδια αλλά δεν δέχθηκαν όλα αυτά να τα βάλουν μέσα σε ένα γενικό πακέτο συμφωνίας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτήν τη δυναμική και ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα δώσει πάτημα στις Κασάνδρες που λένε ότι ήδη πρέπει να τα παρατήσουμε ότι χρειάζεται ένα σχέδιο Β, διότι δεν υπάρχει ένας πλανήτης Β, δεν υπάρχει ένας δεύτερος πλανήτης. Δεν πρέπει λοιπόν να χάσουμε αυτή την ιστορική ευκαιρία που είναι η Κοπεχάγη. Τέλος, εκφράζω την έκπληξή μου. Δεν ανέμενα ποτέ ένας Βρετανός βουλευτής να αμφισβητήσει την αξία του Βρετανικού Κοινοβουλίου που είναι από τις μεγαλύτερες συμβολές της Μεγάλης Βρετανίας στον πολιτισμό. Να είμαστε σαφείς. Η Βρετανική κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε, συνέτυχε στις διαπραγματεύσεις της συνθήκης, ενέκρινε τη συνθήκη, το Βρετανικό Κοινοβούλιο και η Βουλή των Κοινοτήτων και η Βουλή των Λόρδων επικύρωσαν τη συνθήκη η αυτού μεγαλειώτης η βασίλισσα επεκύρωσε τη συνθήκη επομένως το Ηνωμένο Βασίλειο επεκύρωσε τη συνθήκη και ελπίζω όλοι οι Βρετανοί να σέβονται τη λειτουργία του Βρετανικού Δημοκρατικού Συεισετήματος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαρόσο. Τώρα, ο κύριος Ότμαρ Καράς. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Ελπίζω ότι κανένας δεν ε, μισεί σε αυτή την αίθουσα. Ο κύριος Φαράνος μόλις έφυγε. Αλλά ο, το μίσος είναι αντίθετο με το ευρωπαϊκό πνεύμα. Ο εγωισμός, ο εθνικισμός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά δεύτερον στην αίθουσα αυτή ελπίζω να μην υπάρχει κανένας ο οποίος ε, προσπαθεί να φέρει αντιμέτωπο στους πολίτες με την κοινοβουλευτική δημοκρατία και να μην ξεχνάει ότι εμείς είμαστε οι εκπρόσωποι των πολιτών. Όλοι αισθανόσαστε την ένταση πριν από τη διάσκεψη κορυφής. Όλοι περιμένουμε να είναι ε, αποτελεσματική η απόφαση και θετική η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Θέλουμε όλοι να μην <clears throat> παρεμποδιστούμε από ένα άτομο και να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πάρει όλες τις ε, αποφάσεις για προσωπικά και άλλα θέματα. Οι κυβερνήσεις όταν επιλέξουν τους επιτρόπους δεν θα πρέπει να επιλέξουν το μικρότερο κοινό παρανομαστή αλλά την καλύτερη λύση για την κοινότητα της οποίας τμήμα είμαστε. Κάνω έκκληση στις κυβερνήσεις να μην παίξουν στην επιλογή των επιτρόπων τα γνωστά ε, κομματικά παιχνίδια αλλά να θέσουν στο επίκεντρο της επιλογής τους τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητώ από τον πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής φιλόδοξα προφίλ που θα αποστείλει προς τα κράτη-μέλη και στις κυβερνήσεις. Δεύτερο σημείο, εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ε, Ινστιτούτων. Ναι, είμαι υπέρ, αλλά με την μακροεποπτεία δεν θα ε, λύσουμε τα προβλήματα, αλλά χρειαζόμαστε και μια μικροεποπτεία. Δεν χρειαζόμαστε τον μικρότερο κοινό παρανομαστή, χρειαζόμαστε τον μεγαλύτερο κοινό παρανομαστή για να μπορέσουμε να πετύχουμε στους καταλόγους τους Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα. Διακόπτει ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λυπούμε πάρα πολύ, συνάδελφοι. Ο κύριος Γιολάνιν έχει το λόγο τώρα. Ναι, πρόεδρε. Η απέτηση του Βάκλαφ Κλάους για συμπληρωματικά, συμπλήρωμα στην κάρτα ε, βασικών δικαιωμάτων είναι περιττή, αλλά μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί γιατί η κάρτα αυτή αναφέρεται στις πράξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι στο μέλλον. Αν χρειαστεί λοιπόν να σκάνει το Συμβούλιο μια πολιτική δήλωση και να έτσι να πετύχουμε μετά από μερικές εβδομάδες την επικύρωση της ηθίκη που περιμένουμε εδώ και νέα χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να κάνει τις προετοιμασίες, αλλά δεν θα πρέπει να καταλήξει σε γλίγορα συμπεράσματα. Αυτό ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ε, δράση. Ο ύποτος εκπρόσωπος είναι εκείνο που θα πρέπει να δράσει και όχι η δημοκρατία του Συμβουλίου. Ελπίζω η Προεδρία να φροντίσει να μην υπάρχει μονομερή τοποθέτηση της δράσης αυτής, αλλά ένταξή της στο κοινοτικό σύστημα, όπως είπε και ο πρόεδρος παρόσο. Η συνθήκη αυτή μας προσφέρει την, κοινή, την νομική βάση για μια κοινή πολιτική ενέργειας και αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Ελπίζω να διαλυθεί η ομίχλη μέχρι την Κοπεχάγη. Δεν πρέπει να μείνουν τα θέματα αυτά ανοιχτά μέχρι τη διάσκεψη και η Επιτροπή περιβάλλον έθεσε ξεκάθαρα τα θέματα και για τη χρηματοδότηση ελπίζω να συμφωνήσει η διάσκεψη προφή την επόμενη εβδομάδα και χρειαζόμαστε μια εσωτερική κατανομή του κόστου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία και άλλες χώρε θα πρέπει να υποκύψει και θα χρειαζόμαστε καλό καθορισμό των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις αναπτυσσόμενε χώρες. Ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Ντεσαρνέζ. Τρία θέματα θέλω να θίξω. Πρώτον, τι κλιματολογικές αλλαγές. Όλοι το βλέπουν ότι υπάρχει ευθύνη τη Ένωσης ώστε στην Κοπενχάγη να αποτελέσει πρωτοπόρο των χωρών του κόσμου και να διατυπώσει φιλόδοξους στόχους. Ο καθένας μας, ο κάθε χώρα μας πρέπει να κάνει μια χρηματοδοτική προσπάθεια στα μέτρα του. Δεύτερον, το θέμα των μεταναστευτικών ροών. Καλό είναι να λειτουργεί σωστότερα το Frontex. Αν θέλουμε όμως να βοηθήσουμε πραγματικά τις χώρες του Νότου, τότε πρέπει να γίνει εναρμόνιση στο μέτρα δικαιωμάτων ασύλου και ακόμη περισσότερο επιτέλους να υπάρξει μια πραγματική πολιτική της μετανάστευσης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να δούμε τα πράγματα υπεύθυνα και ήρεμα. Τρίτον, για την εξωτερική πολιτική το Συμβούλιο θα αποφασίσει για το θέμα της δημιουργίας αυτής της εξωτερικής υπηρεσίας, θα υπάρξει ο ύπατος αρμοστής ακόμη καλύτερα, αλλά το καλύτερο όλων θα ήταν να μπορούμε να μιλήσουμε με μία φωνή για τις διεθνείς σειράξεις, όπως το Αφγανιστάν. Υπενθυμίζω ότι ο αριθμός Ευρωπαίων στρατιωτών εκεί είναι ισάριθμο σχεδόν με τον Αμερικανών. Έχουν λοιπόν ιδιαίτερη ευθύνη και γι' αυτό οι Ευρωπαίοι. Πρέπει να προτείνουν μια στρατηγική που να μην είναι αποκλειστικά στρατιωτική. Γιατί κανείς άλλος δεν πρόκειται να το κάνει. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Γκέραλντ Χέφνερ. Για δύο ολόκληρα λεπτά. Κυρίε και η τη Λισαβόνα ε, βρίσκεται στην τελική ευθεία και πρέπει τώρα να ταινίσουμε προ τα εμπρό. Θα πρέπει η Ευρώπη να καταστεί πιο κοινωνική, πιο οικονομική, πιο δημοκρατική. ιδίω εκεί έχουμε μεγάλα ελλείμματα. Εγώ θέλω μια Ευρώπη στην οποία οι πολίτε να μην είναι μόνο θεατέ, να μην είναι μόνο αντικείμενο, να είναι υποκείμενα αυτή τη κοινή Ευρώπη. Εγώ θέλω μια Ευρώπη των πολιτών. Και πολλά πρέπει να γίνουν μέχρι να φτάσουμε εκεί. Είπα, ο Λισαβόνα βρίσκεται στην τελική ευθεία και στην τελική ευθεία υπάρχουν πολλά φάουλ. Εγώ δεν έχω καμία κατανόηση ότι τώρα έχουμε έντονες προσβολές του ευρωπαϊκού πνεύματος και του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ένας μόνος από τη της Ευρώπης προσπαθεί να πάρει ο μέρος τους πολίτες του, τη χώρα του, την Ευρώπη. Ότι δεν θα πρέπει να ισχύει η χάρτα ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Και από ό,τι κατάλαβα έγιναν κάποιες υποχωρήσεις. Αυτό θα ήταν απαράδεκτο κυρίες και κύριοι. Θα χαιρόμουν να με διορθώσατε ότι δεν υπάρχει δηλαδή τέτοια διαβεβαίωση γιατί αυτό σήμαινε ότι θα περνάγαμε πάλι στον μεσαίωνα όπου στη μία χώρα ίσχυαν εκείνα τα δικαιώματα που επέτρεπε ο ηγέτης της χώρας αυτής. Αλλά δεν βρισκόμαστε στο μεσαίωνα, βρισκόμαστε σε μία δημοκρατία. Η Τσεχική Βουλή ενέκρινε τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας και είχαν τους λόγους τους, θέλουν η Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ισχύει στην χώρα τους, γιατί είναι η καρδιά της ε, Ευρώπης και θέλουν να βγάλουν από την Ευρώπη την καρδιά της. <clears throat> Τα δικαιώματα των πολιτών δεν είναι διαθέσιμα. Η Ευρώπη δεν είναι ο λογοπάζαρο, είναι μια κοινότητα ανθρώπων δικαίου δημοκρατίας. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε την Κάρτα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, να μην επιτρέψουμε να είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων και καταδεικνούν αυτά που έγινε πόσο σημαντική είναι η Ευρώπη, η δημοκρατία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βλάσεκ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ανταποκριθώ σε αυτά που ελέγχθησαν και να απαντήσω. Είναι σαφές ότι τα θεσμικά όργανα θα βρίσκονται στο επίκεντρο της επόμενης διάσκεψης κορυφής και ιδίω στο θέμα της συνθήκη της Λισαβόνα. Εγώ θεωρώ ότι να συζητάμε το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να γίνεται ταπεινά και με σεβασμό των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στα κράτη-μέλη βάσει των εκάστοτε συνταγμάτων τους. Κάτε με, ένα από τα σημαντικά θέματα της Ιάσης κορυφής θα είναι και η μακροπεριφερειακή πολιτική. Είχαμε συμφωνήσει ότι η Βαλτική είναι ένας καλέας τομέας για την πρόθεση της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για μακροπεριφέρειες και περιμένω ότι θα το επικαιρώσει αυτό η διάσκεψη κορυφής. Πιστεύω επίσης ότι έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου για να σκεφτούμε στην ε, ανάπτυξη της ε, κοινωτικής πολιτικής ε, γιατί αν κοιτάξουμε ένα χάρτη βλέπουμε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στα τέως σύνορα Ανατολής Δύσης. Οι 20 χρόνια μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου εξακολουθούμε να μιλάμε για παλιές και καινούργιες χώρες μέλη. Ευχαριστώ, Λίγο Πρόεδρος. Το χρόνο κύριο Τούσας. ...του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την προσεχή Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σηματοδοτούν ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων στα κράτη-μέλη της με νέα σφοδρή επίθεση ενάντια στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Πρωταρχικό στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κυβερνήσεων των κρατών μελών τη, είτε κεντροδεξιών είτε κεντροαριστερών είναι να διασφαλίσουν τη συνέχιση της κερδοφορίας των μονοπωλίων φορτώνοντας τα βάρη της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ένωση. ενώ η ευρωπαϊκή ένωση ενίσχυσε με πακτολό εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ τα μονοπωλιακά μεγαθύρια χωρίς να αποκλείεται και νέος γύρος χρηματοδότησής τους στη νέα φάση αυτή προκρίνεται γρηγορότερη προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής της λισαβόνας στο επίκεντρο της αντεργατικής επίθεσης βρίσκεται η κατάργηση του οκτάωρου των συλλαγικών συμβάσεων εργασίας και η γενικευμένη εφαρμογή της ευαλφάλειας της προσωρινής ελαστικής και κακοπληρωμένης απασχόλησης με την ενίσχυση του θεσμού των τοπικών συμφώνων απασχόλησης και των stage. στην κλίνη του προκρούστη τίθενται τα δημόσια συστήματα κοινωνική ασφάλισης, υγεία πρόνοιας και εκπαίδευση με σαρωτικέ αλλαγέ σε βάρος των εργαζομένων ανοίγοντας παραπέρα το δρόμο για τη διείσδυση των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων σε αυτούς τους χρυσοφόρους για το κεφάλαιο τομείς. την ίδια περίοδο οι μαζικές απολύσεις πάνω από 5,5 εκατομμύρια τον τελευταίο χρόνο η εργοδοτική τρομοκρατία και η εντατικοποίηση της εργασίας έχουν δημιουργήσει συνθήκες μεσαίωνα στους χώρους δουλειάς χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το διαρκέ έγκλημα που συντελείται σε βάρο των εργαζομένων στην France ε, Telecom, όπου 25 εργαζομένοι έχουν οδηγηθεί στο θάνατο, εξαιτία θάνατο εξαιτία των απαράδεκτων συνδικών εργασίας και τη εντατικοποίησης τη δουλειά Συνάδελφοι, εδώ δεν είναι πράγματα άμα ο καθένας ξεπερνάει κατά μισό λεπτό Και μένα με δυσαρεστεί αυτό που αναγκάζομαι να σας διακόπτω. Θέλω να τηρείτε το χρόνο ομιλία σας ο καθένας, αλλιώς δεν μπορεί να γίνει συζήτηση. Λοιπόν, επόμενος ομιλητής, Γουλιέλμος ο κόμις του Ντάρτμο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το μεγάλο πρόβλημα για τα κράτη-μέλη είναι όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος Μπίσκι η κρίση της απασχόλησης. Η ανεργία των νέων είναι 24% στη Γαλλία, 25% στην Ιταλία, 39% στην Ισπανία. Και όμως μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα ασχοληθεί μόνον με, άλλες, με θριαμβολογίες για την επιτυχία δήθεν των μέτρων αντιμετώπισης και για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Όλες οι κινήσεις προς τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού υπερκράτους τελικά έγιναν με χειραγώγηση και τόσο αδιάντροπα ώστε η συνθήκη δεν έχει καθόλου δημοκρατική νομιμότητα και αυτό θα έχει συνέπειες. Ήδη φαίνεται και το καταλαβαίνουν όλοι. Trzymanie się w czasie, to bardzo ważne. E, pan Czanat Segedi. Ο κύριο Σέγγεντι τώρα, για 1,5 λεπτό. Κυρία, ε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Προεδρεύουσα, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκίνησε μια συζήτηση εντελώς επιφανειακή για τη συνθήκη της Λισαβόνα γιατί δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τίποτα μεταξύ μας. Να μιλήσουμε για μια μειονότητα στην Ευρώπη που δεν έχει κανένα δικαίωμα. Ένας Ούγγρος που κατοικεί από την άλλη μεριά των Καρπαθίων. Έχουμε εκατομμύρια Ούγγρους οι οποίοι δεν χαίρουν κανενός δικαιώματος στη δική τους επικράτεια. Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι που κατοικούν στη Ρουμανία δεν μπορούν να μιλήσουν τη γλώσσα τους, δεν μπορούν να την μελετήσουν, δεν μπορούν να ασκήσουν τη θρησκεία τους. Υπάρχει και ένα διάταγμα που απαγορεύει τη χρήση της Ουγγρικής γλώσσας και υπάρχουν πολιτικοί που χρησιμοποιούν ω διαπραγματευτική εντολή το διάταγμα Μπένες. Αυτό είναι δικτατορία, είναι ρατσισμό να θεωρεί κανείς το διάταγμα Μπένες ω διαπραγματευτικό χαρτί. Κρυβόμαστε πίσω από τη δημοκρατία για να καλύψουμε τη δικτατορία. Θέλουμε μια δημοκρατική Ευρώπη, χωρίς συνθήκη της Λισαβόνας, χωρίς διατάγματα Μπένες, χωρίς διακρίσεις των Ούγγρων. λέγεται ότι δεν ισχύουν οι συνθήκες, ε, το διάταγμα του Μπένες. Αλλά πότε θα αποζημιωθούν οι Ούγγροι των Καρπαθίων. Σε αυτό το κοινοβούλιο που ασχέτως του θέματος που συζητείτε πάντα το ίδιο θέμα συζητούν. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να βρεθεί μία λύση, ούτω ώστε η τσεχική δημοκρατία να ολοκληρώνει την επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας. Πρέπει να είναι δίκαιη ε, αυτή η επικύρωση, είναι απόδοση συγγνώμη, δικαιοσύνης προς όλα τα κράτη-μέλη. Η οικονομική κρίση έχει υποσκάψει σημαντικά τα δημοσιονομικά των χωρών. 24 κράτη παρακολουθούνται σήμερα από κοντά από την Κομισιόν λόγω του σημαντικού ελλείμματος. Όσοι είχαν δεσμευτεί με το σύμφωνο σταθερότητας έχουν πρόβλημα σήμερα λόγω της κρίσης και των υψηλών δημοσίων δαπανών. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες της κάθε χώρας και θα πρέπει να βοηθήσουμε σε μία συμφωνία για την στρατηγική εξόδου από την κρίση και την έγκριση διαρθρωτικών μέσων για την λήψη διαρθρωτικών μέτρων για να βγούμε από την κρίση και να σταθεροποιήσουμε την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε με τις δημόσιες ενισχύσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάλουσες συνθήκες στα κράτη-μέλη. Η κυρία Λίζα Γιάκονσάρη. Συμφωνώ κύριε Πρόεδρε με την κυρία Μαρινέσκου. Το Συμβούλιο πρέπει να βρει κάποια λύση και γρήγορα για να είμαστε και εμείς σε θέση να αρχίσουμε επιτέλους να εφαρμόζουμε τις συνθήκες Λισαβόνας και να βγούμε από την κρίση. Κρίση που πλήττει σκληρά την Ευρώπη και πρέπει ο κόσμος να μπορέσει επιτέλους να επιστρέψει σε μια πληρέστερη απασχόληση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντέδρασε και γρήγορα για να αναγκάσει τις Ηνωμένε Πολιτείες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Θα ήταν περίεργο λοιπόν να έχουμε τώρα την εντύπωση ότι η κρίση δεν πέρασε. Γιατί αυτό συμβαίνει. Υπάρχουν ακόμη σημαντικά προβλήματα όπως η γύρανση του πληθυσμού, η ανεργία, η ανάγκη της αναδιάρθρωσης των αυτοκινητοβιομηχανιών και στην καρδιά της κρίσης αυτής υπάρχει το γεγονός ότι εμείς οι πολιτικοί πρέπει να δείξουμε, να βρούμε κάποια λύση. Η Κομισιόν προσπαθεί να διαρθρώσει τα θεσμικά και ελπίζω και το Κοινοβούλιο να μπορέσει να συμβάλλει στην εξέβρεση της λύσης αυτής. Ευχαριστώ κυρία Σιλβάνα Κοχμερίν έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Κομισιόν, κύριε Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, θα προτιμούσατε φαντάζομαι να έχετε δύο εβδομάδε στη διάθεσή σα για διάσκεψη κορυφή και όχι δύο μέρε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά θέματα που πρέπει να εξετάσετε. Έχουμε τα πιο σημαντικά για του πολίτε, την οικονομική κρίση και την υπέρβαση σε προοπτικέ για απασχόληση, κλιματολογικέ αλλαγέ και το Αφγανιστάν. Τα θέματα αυτά δεν είναι νέα. Αυτό που είναι νέο είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι δυνατόν να συζητηθούν όλα τα θέματα αυτά με προοπτική να μπορέσει να καθιστεί ικανή προεργασία ή προσεργασία συγγνώμη, η Ευρώπη με τη νέα συνθήκη. Θα πρέπει να δράσετε αποτελεσματικά όσον αφορά και την, εξωτερική, ε, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, και όσον αφορά και την προετοιμασία της διάσκεψης προφήσης στην Καμενχάγη και σχετικά με την μελλοντική δομή ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και εκεί θα πρέπει να δράσετε. Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι ε, δηλώσει επιτυχίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα εύχομαι κάθε επιτυχία και καλή τύχη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι δεν μπορώ να μιλήσω καταλανικά διότι παρόλο που είναι μία γλώσσα πάνω από 10 εκατομμύρια, τη μιλούν πάνω από 10 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν μπορώ να μιλήσω καταλανικά και θα μιλήσω Ιταλικά. Η Φιλανδία αναγνώρισε το δικαίωμα σε όλους τους πολίτες να έχουν σύνδεση με το ίντερνετ ως γενικό δικαίωμα διότι επιτρέπεται έτσι το, η πρόσβαση πρόσβαση στο δικαίωμα της γνώσης έτσι όπως ορίζεται αυτό το δικαίωμα και από τη συνθήκη της Λισαβόνας για το δικαίωμα δηλαδή, της πληροφόρησης και της γνώσης. Θα κάνει κάτι το Συμβούλιο ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ένα παγκόσμιο παράδειγμα και προς αυτή την κατεύθυνση. Μάρτιν Κάλενεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολλά σημαντικά θέματα θα συζητηθούν από το Συμβούλιο, αλλά κατ' εμέ ένα από τα σημαντικότερα είναι το μέλλον της συνθήκης της Λισαβόνας. Εδώ πολλοί ομιλητές και ομιλήτριες αναφέρθηκαν στο ότι η συνθήκη λέει θα αυξήσει το δημοκρατικό χαρακτήρα στη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών και δεν αστείευονταν. Παρόλα αυτά δεν βλέπουμε κανέναν τέτοιο δημοκρατικό χαρακτήρα εφόσον έγινε προσπάθεια εξαπάτησης των λαών εφόσον αποφεύθηκαν τα δημοψηφίσματα. Τα σχόλια του κυρίου Μπαρόσου προηγουμένως ήταν ενδιαφέροντα. Θα σας εξηγήσω γιατί οι Βρετανοί είναι ακόμη θυμωμένοι. Και τα τρία πολιτικά κόμματα στις προηγούμενες εκλογές είχαν δεσμευτεί να γίνει δημοψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα όπως λεγόταν τότε αν και άλλαξε όνομα. Και δύο από αυτά τα κόμματα τελικά υπαναχώρησαν και αρνήθηκαν το δημοψήφισμα. Άρα είναι θέμα δημοκρατίας. Πού είναι ο δημοκρατικός χαρακτήρας. Αν δεν είχε υπάρξει αυτή η υπόσχεση τότε θα είχε δίκιο ο κύριος Μπαρόσο ότι θα είχε υπάρξει δημοκρατική διαδικασία επικύρωσης. Δεν χρειάζεται να μας δίνει μαθήματα ο κύριος Μπαρόσο εδώ μέσα εφόσον υποστηρίζει εκείνους που αρνούνται στον κόσμο το δικαίωμα στο δημοψήφισμα. Γι' αυτό οι περισσότεροι Βρετανοί είναι τόσο αρνητικοί. Στην Ιρλανδία ζήτησαν δύο φορές δημοψήφισμα. Σε εμά ούτε μία. Δεν ξέρω λοιπόν πώς μπορεί κανείς να μιλάει για αυξημένο δημοκρατικό χαρακτήρα εφόσον δεν δίνεται κανένας λόγος στους περισσότερους λαούς της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Μάριο Μποργέζιο, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να κάνω εδώ ορισμένες παρατηρήσεις ε, σχετικά ε, με την μελλοντική ισχύ της συνθήκης ε, της Λισαβόνας. Και αυτό δηλαδή και λόγω της απόφασης του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου για τη Λισαβόνα. Θέλω να μην πω ότι δεν υπάρχει ε, δημοκρατική νομιμότητα λόγω της ανεπαρκούς εκπροσώπησης ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των χωρών με τον περισσότερο πληθυσμό αλλά και λόγω της ανεπαρκούς ε, παροχής εξουσίας και αρμοδιοτήτων στα εθνικά κοινοβούλια για την άσκηση των ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων. Αλλά και κάτι άλλο, ένα τρίτο στοιχείο, δεν αναγνωρίζεται καθόλου τα περιφερειακά κοινοβούλια η αρχή της επικουρικότητας θάβεται πλήρως από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου θα έπρεπε να είχε ανοίξει με μια μεγάλη νομικοπολιτική συζήτηση σε αυτό το κοινοβούλιο και αυτό λόγω των κινδύνων που ενηχεύει αυτό το σχέδιο μοσπονδιοποίησης της Ευρώπης. Και θέλω να θυμίσω εδώ και τα δικαιώματα των εθνών χωρίς κράτος από την χώρα του Πάδου στην Βρετάνη, στην ε, ε, ε, πρέπει να τα θυμίσουμε όλα αυτά, διότι αυτό που θέλανε οι πατέρες της Ευρώπης να οικοδομήσουν ήταν η Ευρώπη των λαών και όχι η Ευρώπη των μεγάλων συμφερόντων. Ευχαριστώ κύριε Μποργέτσιο. Το λόγο έχει ο κύριος Φρανς Ομπερμάιερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα της παράνομης βασταμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να σας τονίσω ότι στο περασμένο χρόνο αυξήθηκε σημαντικά. Όπως είπε η Κομισιόν, αυξήθηκε κατά 63% η παράνομη μετανάστευση. 2008 υπήρχαν ε, ε, τεράστια αριθμοί ε, παρανόμων λοιπόν. Στη Αυστρία λόγω της γεωγραφικής θέσης είναι ένας πολύ αγαπητός ε, ε, στόχος. Παραδείγματος χάρη 48 Κούρδοι ζήτησαν ε, άσυλο ο αριθμός όσο πάει σε μία μέρα όσο πάει αυξάνεται ο αριθμός αυτός και απειλούνται οι ίδιοι οι πολίτες μας και κάνω έκλειση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 29 και 30 του Οκτωβρίου να λάβει υπόψη και αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπρόκ. Δύο λεπτά. Πρόεδρε, Κυρία Αντιπρόεδρε της Κομισιόν, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Θεωρώ ότι η συνθήκη της Λισαβόνα θα πρέπει τώρα γρήγορα να στρεφεί σε ισχύ και να εφαρμοστεί. Εδώ και δέκα χρόνια συζητάμε ε, θεσμικά το θέμα αυτό. Φτάνει. Πρέπει τώρα κάτι να κάνουμε για τους πολίτες, Ιδίω τη σημερινή στιγμή της οικονομικής κρίσης, να βοηθήσουμε τους πολίτες στην καταπολέμηση της ανεργίας κλπ. Γι' αυτό παρακαλώ και τον πρόεδρο Κλάους να ανοίξει τη οδό τώρα αφού έχει επικυρωθεί η συνθήκη αυτή ε, σε 27 χώρες και στην Τσεχική Δημοκρατία δύο φορές το δημοτικό Δικαστήριο είπε εντάξει. Τι τρίτη θα το ξανακάνει. Λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο το εθνικό δίκαιο δεν ακυρώνεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θα πρέπει να το πούμε αυτό ξεκάθαρα. Θα μπορούσε να κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενδεχομένω με σχετική δήλωση, αν χρειαστεί, α το κάνει. Αλλά δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο για καμία χώρα. Θα ήθελα να σα πω ότι η συνθήκη αυτή για κατά την εφαρμογή του θα πρέπει να αναφέρεται στι βασικέ αρχέ. Αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, δημοκρατία. Αυτό θα συζητήσουμε και σήμερα το απόγευμα. Αναφέρομαι εδώ συγκεκριμένα στην υπηρεσία εξωτερική δράση. Η, ιδέα τη αποτελεσματικότητα δεν θα πρέπει να ακολουθεί ει βάρο της διαφάνειας και τη δημοκρατικότητα και των δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ούτε ει βάρο τη αρχή της κοινοτικότητα. Θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητε διασφαλίσει. Και γι' αυτό, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, θα ήθελα να σας παρακαλέσω κάποιες ολοδοξίες που έχει η κυβέρνησή σας να τις εγκαταλείψετε. Δηλαδή ήδη την επόμενη εβδομάδα να αποφασίσετε η διάσκεψη κορυφής κατευθύνες γραμμές για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Όχι. Καλύτερα να περιμένετε και να υπάρχει μια κοινή απόφαση με τον ύπατο εκπρόσωπο και να υπάρχει μια δίκαια βάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπρόκ. Ο κύριος Δέρτμον θέλει να σας ρωτήσει κάτι με την μπλε κάρτα. Κύριε Μπρόκ, το δέχεστε, ναι, για 30 δευτερόλεπτα. Κύριε Μπρόκ, είπατε ότι επί 10 χρόνια συζητιέται η συνθήκη της Λισαβόνας. Έχετε όμως καταλάβει ότι εσείς και οι συνάδελφοί σας δεν έχετε πείσει εδώ και 10 χρόνια τον κόσμο για την αξία της και ότι χρειάστηκε να κάνετε αυτές τις χειραγωγήσεις τις κατάπτυστες για να επικυρωθεί η συνθήκη. 30 δευτερόλεπτα ο κύριος Μπρόκε να απαντήσει. Ε, κύριε συνάδελφε, οι θεσμικοί εισαλλαγές της νοικίας έτυχε πάνω της ευρείας ε, υποστηρίξη του ευρωπαϊκού λαού και των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών. Πάντα κάποιες μεμονωμένες χώρες αποφάσισαν διαφορετικά για λόγους ιδίως εσωτερικής πολιτικής. Τώρα 27 κράτη αποφασιστήκαν κοινοβουλευτικά, μια δημοκρατική απόφαση κοινοβουλευτισμό δεν είναι ε, δημοκρατία δεύτερης κατηγορίας. αποφάσισα λοιπόν κοινοβουλευτικά ή με δημοψήφισμα. Και γι' αυτό η συνθήκη της Λισαβόνα εγκρίνεται από τη μεγαλύτερη πλειοψηφία του πληθυσμού και της δική σα χώρα. Ευχαριστώ κύριε Μπρόκ για 1,5 λεπτό ο κύριος Ρούσεκ. Θα ήθελα να κάνω και εγώ μερικά σχόλια ως προς την επικύρωση της συνθήκης στην Τσεχία. Οι Τσέχοι μέσω των εκλεγμένων εκπροσώπων τους έχουν σαφώς δεχτεί τη συνθήκη της Λισαβόνας. Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, οι Τσέχοι θέλουν ο πρόεδρος Κλάους να, να επικυρώσει τη συνθήκη και μάλιστα σύντομα. Και τρίτον, επίσης οι Τσέχοι θέλουν να υπάρχει να υπάρχει εγγύηση των ε, δικαιωμάτων τους ισότιμα με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Δηλαδή δέχονται και τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνεται στη συνθήκη. Ο πρόεδρος Κλάους είναι γνωστός για την αντίστασή του κατά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και τώρα χρησιμοποιεί προφάσεις για να δοθούν πρόσθετες εγγυήσεις στη τσεχική δημοκρατία. Η Ένωση δεν πρέπει να δεχτεί το παιχνίδι αυτό του κυρίου Κλάους. Πρέπει η πλήρης συνθήκη να επικυρωθεί χωρίς εξαιρέσεις και με την κοινωνική της πτυχή. Είναι ντροπή που ο πρόεδρός μας 60 χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου προσπαθεί να ξαναθέσει θέμα Σουδιτών, οι οποίοι υπέφεραν τόσο πολύ κατά τον πόλεμο αλλά και μετά. Είμαι σίγουρος ότι εκείνοι έχουν πάρει μαθήματα από τη στρατηγική του και γνωρίζω ότι και οι Σουδίτες και οι Τσέχοι και οι υπόλοιποι Γερμανοί θέλουν να ζήσουν ειρηνικά και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρούσεκ. Η Φιώνα Χόλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Σουηδική Προεδρία είπε ότι είναι πολύ σημαντική χρηματοδότηση των μέτρων αντιμετώπισης των κλιματολογικών αλλαγών. Συμφωνώ. Αλλά η προσφορά της Κομισιόν, η πρότασή της είναι τελείως ανεπαρκής. Ιδίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο κ. Μαρόσο είπε προηγουμένως τα 100 δισεκατομμύρια το χρόνο που χρειάζονται για τις αναδυόμενες ε, χώρες για να αντιμετωπίσουν κλιματικές αλλαγές θα καλυφθούν από τις συναλλαγές των εκπομπών. Δεν υπάρχει όμως καμία βεβαιότητα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε δει πόσο ασταθείς είναι οι τιμές του διοξιδίου και πόσος καιρός θα χρειαστεί για να γίνουν οι συναλλαγές αυτές. Τρίτον, οι αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες θεωρείται ότι εύκολα θα χρηματοδοτήσουν τα μέτρα αντιμετώπισης. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αφού και οι ίδιοι έχουμε δυσκολίες για να τα χρηματοδοτήσουμε. Γιατί θεωρούμε ότι οι αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες μπορούν, χρειάζεται πρόσθετα κονδύλια για όλα αυτά. Ευχαριστούμε. Ανδρέας Μόλτσερ. Πρόεδρε, επιτρέπω να κάνω τρεις παρατηρήσεις για τη διάσκεψη κορυφής. Καταρχήν, το Ολλανδικό ναι βασίζεται κυρίως στην οικονομική κρίση. Πριν από ένα χρόνο δόθηκαν δισεκατομμύρια ε, για να διασωθούν οι τράπεζες. Τώρα έχουν πάντα πάλι οι τραπεζίτες όμως εισοδήματα ρεκόρ. Πώς συμβάζω αυτά. Δεύτερον, χάρη στη θήκη της Λισαβόνας υπάρχουν τώρα νέες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό... Οι υποψήφοι αυτοί είναι συνήθως παλιοί πολιτικοί που έχουν αποτύχει δημοκρατικά στις χώρες τους. Ο πρόεδρος της ε, Επιτροπής ε, του Συμβουλίου ή ο ύπατος εκπρόσωπος ε, αν εκλεγούν κατά τέτοιο τρόπο θα έχουμε ένα χάος. Επίσης λέγεται ότι θα πρέπει να πάρει μία υποσημείωση ο Βακλαφλάος όσον αφορά τα διατάγματα πένες για να μπορέσει να υπογράψει. Τότε υπάρχουν διαφορετικά βασικά δικαιώματα για τους Γερμανούς, για τους Σουδίτες και για τους άλλους. Δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ο Σάριος Βόλσκι. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας Αναμένουμε να γίνει πρόοδος στο Συμβούλιο και για το κύριο θέμα της υπηρεσίας εξωτερικών για να δημιουργηθεί επιτέλους μία κοινή ευρωπαϊκή διπλωματία για να υπάρχει συνέπεια στις εξωτερικές δράσεις που πρέπει να αναλάβουμε αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε εξωτερικές απειλές και προβλήματα όπως τη διασφάλιση των ενεργειακών προμηθειών μας. Αναμένουμε λοιπόν από το Συμβούλιο να λάβει υπόψη του τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενεκρίθη αυτή την εβδομάδα στη Θεσμική Επιτροπή για να υπάρξει πραγματική εξωτερική πολιτική πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα εργαλεία ώστε ο μελλοντικός ύπατος αρμοστής της να είναι σε θέση να πάρει τα μέτρα που πρέπει να πάρει σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες του πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τη διεύρυνση, την πολιτική γειτονία, την ε, εμπόριο κλπ. Το κύριο θέμα εδώ που τίθεται είναι η δημοκρατική νομιμότητα που μπορεί να υπάρξει μόνο εάν συνεργαστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. το οποίο πρέπει να τύχει διαβούλευση κατά, κατά το καθορισμό ήδη των στόχων και των δικαιοδοσιών της υπηρεσίας αυτής και αφότου αρχίσει να λειτουργεί πρέπει το Κοινοβούλιο να παίζει σημαντικό ρόλο και στην εξέταση και εφαρμογή των προγραμμάτων που θα έχει εγκρίνει η υπηρεσία αυτή. Η δημοκρατική νομιμότητα της νέας αυτής υπηρεσίας θα εξαρτηθεί και από τη σύνθεσή της, τη γεωγραφική εξισορρόπηση την ισότιμη μεταχείριση όλων των χωρών που είναι μία από τις βασικές αρχές μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Άριους Βόλσκι και τώρα για 1,5 λεπτό η κυρία Περβάν Συμπερές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Μετά από τέσσερις μήνες από τις εκλογές, ευρωεκλογές Ακόμη δεν έχει αρχίσει η κανονική λειτουργία της Ένωσης εν ώψη της Λεσαβόνας. Εδώ τίθενται τα εξής προβλήματα. Πρώτον, ένα χρόνο μετά την εκπεφρασμένη αλληλεγγύη όλων των χωρών μελών προς τις τράπεζες πρέπει επιτέλους να αναλάβετε την πρωτοβουλία επιβολής ενός φόρου για τις χρηματικές συναλλαγές ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν όντως να ασκήσουν κάποια αλληλεγγύη. Έπειτα, εξ ονόματος της Κομισιόν, ο πρόεδρος της εχθές μας είπε ότι υποστήριζε τον προϋπολογισμό όπως έχει σήμερα. Ένα χρόνο δηλαδή μετά το πρόγραμμα αναθέρμανσης δεν έχει φανταστεί τίποτε πιο καινούριο. Ε, τι έχουμε δει το τελευταίο αυτό χρόνο, ότι η ανεργία συνεχίζεται και αυξάνεται ο προϋπολογισμός που έχουμε μπροστά μας σήμερα δεν χρηματοδοτεί καθόλου ούτε καν το δεύτερο μέρος του σχεδίου αναθέρμανσης που σκέφτηκαν πέρυσι. Πρέπει λοιπόν και επ' αυτού να κινητοποιηθεί το Συμβούλιο. Φορολόγηση των χρηματικών συναλλαγών, αλληλεγγύη και ένα πραγματικό σχέδιο αναθέρμανσης και στο δεύτερο μέρος του να εφαρμοστεί. Ευχαριστούμε κυρία Μπέρε. Το λόγο έχει τώρα για ένα λεπτό η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι που βλέπω την πρώην συνάδελφό μας Μάλστρομ μπροστά μας σήμερα. Το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία με τη θετική του εξέλιξη και η μελλοντική έγκριση από τον πρόεδρο της Πολωνίας είναι ενθαρρυντικά, ενθαρρυντικές εξελίξεις. Το θέμα όμως είναι να δούμε τι θα κάνουμε γενικά με την κρίση. Αυτό ε, αφορά τους πολίτες και όχι η Λισαβόνα. 27 εκατομμύρια ψήφισαν υπέρ, 24 λένε κατά. Αυτή είναι η δημοκρατική νομιμότητα που έχουμε. Πρέπει όμως επιτέλους όλα αυτά να καταλήξουν σε μια νέα ορμή. Εκατό εκατομμύρια ευρώ και πεντακόσια σε είναι θετικά μέτρα αλλά δεν αρκούν για να μπορέσει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα που είναι οι επενδύσεις. Ευχαριστούμε κυρία Χάρκιν. Τώρα για δύο λεπτά. Βάντεν Κάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε. Είναι πολύ καλό η Ευρώπη να επωφεληθεί από την επιτυχία του Ιρλανδικού δημοψηφίσματος. Έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τη συνθήκη της Λισαβόνας. Όλοι ανησυχούμε για τους Τσέχους και θα περιμένουμε με σεβασμό την απόφαση του δικαστηρίου τους, αλλά σας παρακαλώ να είστε υπομονετικοί με τον κύριο Βάκλαβ Κλάους, διότι αν τον πιέσουμε αυτό μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό. Δεύτερο σημείο, η Κοπενχάγη και η επιτυχία της αποτελεί πηγή ελπίδας για την Ευρώπη και για τον κόσμο. Η αηφορία βρίσκεται στην πηγή της τεχνολογικής πρόοδου. Έχουμε σήμερα σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις που επιτρέπουν την καταπολέμηση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κρίσης ταυτόχρονα. Τώρα για να πάω στην κρίση. Χρειάζεται προστασία των θέσεων απασχόλησης. Τα σχέδια του Συμβουλίου είναι καλά, αλλά για πολλούς πολίτες ε, τα σχέδια του Συμβουλίου είναι άγνωστα. Η ρύθμιση του τραπεζικού τομέα είναι θεμελιώδης και ελπίζω ότι θα προχωρήσετε και προς αυτό το τομέα την επόμενη εβδομάδα για να τελειώνω. Το θέμα του ασύλου Υποστηρίζω όλες τις προθέσεις της Σουηδικής Προεδρίας. Όταν δεν ε, έχουμε όμως αποτελέσματα από το Συμβούλιο υπάρχει πρόβλημα και ακούστηκε και στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθερών αυτό το πρόβλημα ότι δεν έχουμε καταλήξει σε λύσεις. Ο Τζανλούκα Σούστα τώρα για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάψει αυτή η Ολομέλεια να συζητάει επάπειρον για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει να, γίνουνε να γίνει σεβαστή η βούληση αυτού του Κοινοβουλίου των, και των 26 που ψήφισαν δημοκρατικά, έστω και με διαφορετικές μορφές αυτή τη συνθήκη. Οι προσβολές προς τη συνθήκη και το δημοκρατικό της περιεχόμενο πρέπει να απορριφθούν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας είναι μία σημαντική ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της Ευρώπης, όχι μόνο την οικονομική κρίση αλλά και το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών. Αυτά που μας είπαν μέχρι σήμερα προδρεύοντες είναι ανεπαρκή διότι δεν γίνεται μια σημαντική, ε, μια δυναμική ερμηνεία της νέας συνθήκης και δεν καλύπτεται αυτό το οποίο προβλέπεται στην ατζέντα της Λισαβόνας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υποβολή προτάσεων από την Κομισιόν για την καταπολέμηση της κρίσης, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την απασχόληση και το Συμβούλιο θα πρέπει να απαντήσει σε αυτές τις οικονομικές προκλήσεις άμα θέλουμε εμείς να παραμείνουμε μια μεγάλη οικονομική δύναμη ο Ήπειρος. Λείπει που θα γίνουμε και μια υπερδύναμη σε εξωτερικά επίπεδα. Λείπει λοιπόν ένα πρόβλημα ανάκαμψης, λείπει μια ευρωπαϊκή πνοή με ένα με ψηλό προφίλ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά περιμένουμε από το επόμενο Συμβούλιο στα τέλη του μηνός. Ευχαριστώ κύριε Σούστα. Ο Γιώχαν Κορνέλης Βαν Μπάλεν. Είναι πολύ σημαντικό κύριε Πρόεδρε να καταπολεμήσουμε την οικονομική κρίση Άρα να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να ακολουθήσουμε τις συστάσεις της Επιτροπής στο Ιντερκ και η Κομισιόν και το Συμβούλιο να δεσμευτούν γιατί πρέπει να μειωθεί οπωσδήποτε η γραφειοκρατία. Έπειτα το πρωτόκολλο της Άγκυρας. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είπε σε μία διάσκεψη στη Χάγη ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να επικυρώσει και άρα να εφαρμόσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας. Αυτό είναι επίσημη δήλωση της 7ης Οκτωβρίου. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν απλώς να ξαναζητήσουμε. Η 1η Νοεμβρίου είναι διορία που πρέπει να τη σεβαστούμε. Τι θα κάνουμε, ρωτάω. Ευχαριστούμε κύριε Βανμπάλεν και τώρα για δύο λεπτά ο κύριος Χόκμαρκ. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία σας εδώ και θα ήθελα να σχολιάσω την τελευταία σύνοδο του Συμβουλίου. Καταρχήν για τις κλιματολογικές αλλαγές είναι σημαντικό να πάμε στη διαπραγμάτευση προσπαθώντας να, με στόχο την καλύτερη δυνατή λύση. Και η καλύτερη δυνατή λύση δεν πρόκειται να επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή όλων. Το λέω γιατί καμιά φορά συζητάμε. Λες και η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη της ήταν ικανή να εφαρμόσει την καλύτερη δυνατή λύση. Ενώ υπάρχει και η Κίνα και η Ινδία και άλλες χώρες που πρέπει να συμμετάσχουν στις προσπάθειες αυτές κατά πολέμηση των επιπτώσεων των κλιματολογικών ελεγχών. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε ρεαλιστικά. Και γι' αυτό όλες οι χώρες να είναι διατεθειμένες να αναλάβουν δεσμεύσεις. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να δεχτούμε οι δεσμεύσεις τρίτων χωρών να εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις μόνον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, χρειάζονται υγιή προγράμματα παντού. Δεύτερο θέμα, κύριε Πρόεδρε, οι χρηματοπιστωτικές αγορές πρέπει να είναι σταθερές. Και αυτό δεν σημαίνει απλώς σταθερότητα της μακροοικονομίας, πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της διευθέτησης των πλεονασμάτων. Και αυτό ξεπερνάει κατά πολύ την απλή επίλυση της τωρινής χρηματοπιστωτικής κρίσης. Χρειάζεται σταθερότητα των αγορών, αλλά γι' αυτό χρειάζεται και σταθερές επενδύσεις και σταθερή ανάπτυξη και σταθερή απασχόληση. Και άρα όλα τα νομοθετικά μέτρα που πρέπει να πάρουμε να λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις μεταβλητές και τις παραμέτρους. Δεν αρκεί να επενδύουμε σε ορισμένες μόνο χώρες γιατί έτσι αποσταθεροποιούμε τις δικές μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μάρκ. Και τώρα για 1,5 λεπτό ο κύριος Χουάν Λόπες Αγγιλάρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μόλις έγινε το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία όπου κάνει πιο πιθανή τη θέση σε ισχύ της συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα έχουμε τα θεσμικά όργανα τα οποία θα μπορούν να ασχοληθούν με τα ζητήματα που μας απασχολούν, την δημιουργία θέσεων εργασίας, τις κλιματικές αλλαγές, τις ενεργειακές μας ανάγκες, το δίκαιο εμπόριο. Και οι ψηφιακέ ε, ανάγκες θα τεθούν επιτάπητος. Είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία για να δώσουμε μια όθηση στις προτεραιότητες της νέας επιτροπής, ε, κατά την άποψη του κ. Μπαρόζο τουλάχιστον. Αυτό το λέω ως μέλος της ομάδας των σοσιαλιστών. Αυτό που θέλουμε είναι μια ισόρροπη σύνδεση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό και ο ύπατο εκπρόσωπο να προέρχεται από τη δική μα πολιτική οικογένεια. Αλλά κυρίω πρέπει να υπάρχει και ε, ισοτιμία μεταξύ των φίλων, ισότητα μεταξύ των φίλων στα μέλη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει τα σωστά χαρτοφυλάκια να τα αναλάβουν τα κατάλληλα άτομα. Και αυτό το λέω στα πλαίσια τη γενική συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να έχουμε μια επιτροπή που να είναι υπεύθυνη για τη δικαιοσύνη και. Μάλλον μια επίτροπο, έναν επίτροπο υπεύθυνο για τη δικαιοσύνη και τι εσωτερικέ υποθέσει. Και έναν άλλον για την ασφάλεια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να υπόκειται στην ε, ασφάλεια, να αποτελεί μέρος της. Θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα διαφορετικό επίτροπο για τη μετανάστευση, ότι υπάρχει μια σαφή ε, διάκριση μεταξύ των διαφορετικών αρμοδιοτήτων και να έχουμε υπόψη μας πάντα και τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό ο κύριος Κρόουλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επίτροπο. Όταν συζητούμε για τι συνόδου αυτέ, μα έρχονται πολλέ ιδέε. Σα θυμηθούμε πριν από 10 χρόνια παρόμοιε προτάσει που προέρχονταν από μέλη του Κοινοβουλίου, μέλη του Συμβουλίου και επίση από διάφορου επιτρόπου. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει αποδειχθεί είναι ότι δεν πετυχαίνουμε πάντα του στόχου μα. Αλλά σίγουρα κάτι το πετυχαίνουμε, ότι η Ένωση λειτουργεί βάσει τη αλληλεγγύη, με μεγάλα σχέδια και μεγάλου στόχου και μεγάλε φιλοδοξίε. Και έτσι κινείται ο κόσμο μα. Πρέπει πάντοτε να έχουμε μεγαλύτερα σχέδια και μεγαλύτερε φιλοδοξίε για το μέλλον. Πολλοί μίλησαν για την αύξηση της ανεργίας, κάτι που πλήττει τόσα τόσου πολίτε ε, τον τελευταίο καιρό. Όμως, εδώ πρέπει να ληφθεί, αναλυφθεί σοβαρή δράση για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Τα προβλήματα της ρύθμισης και το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόνται πολλές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν δημιουργήσει. Πρέπει λοιπόν η πολιτική μα να λαμβάνει υπόψη την αλληλεγγύη. Γιατί όταν μιλάμε για αλληλεγγύη, δεν θέλουμε οι μεγάλοι να στρέφονται κατά των μικρών. Το G20 είναι κάτι που θα μπορούσε και αρνητικά να επηρεάσει τι μικρέ χώρε και τι μεσαίε χώρε, οι οποίε αναδύονται αυτή τη στιγμή οικονομικά. Επίση, ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να μα απασχολήσει είναι τα πνευματικά δικαιώματα Σίγουρα αυτό έχει συζητηθεί στη Σουηδική Προεδρία και έχει να κάνει με όλε αυτέ τι ε, ανησυχίε. Ευχαριστούμε κύριε Κρόουλη. Και τώρα για δύο λεπτά ο κύριο Κέλλαμ. Πρόεδρε, Υπουργέ, Επίτροπε. Η συνθήκη τη Λισαβόνα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ και άρα ζούμε μια ιστορική στιγμή. Και πρέπει να επικεντρωθούμε πρώτα απ' όλα στο κοινό μέλλον τη Ευρώπη και στο κοινό καλό φοβάμαι ότι δεν είναι η βέλτιστη ευκαιρία. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε αυτέ τι τελευταίε στιγμέ για να προάγουμε εθνικά συμφέροντα. Οι παγκόσμιε προκλήσει για την Ευρώπη δεν μπορούν να ρυθμιστούν χωρί αποτελεσματικά κοινά θεσμικά όργανα και κοινέ πολιτικέ. Όμως σήμερα ε, χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ ηθική δέσμευση και μια κοινή αντίληψη σχετικά με τις ευρωπαϊκές αξίες ε, όπως αυτές που μας πρότειναν οι πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταπολεμήσουμε τον εθνικό εγωισμό. Και γι' αυτό για την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε μόνο ε, ε, καλή πορεία των επιχειρήσεων. Χρειαζόμαστε ένα όραμα, χρειαζόμαστε κύρος, ούτως ώστε να επιφέρουμε αλλαγές ε, στην Ευρώπη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε σαφή δέσμευση και ουσιαστική εφαρμογή των πολιτικών από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν χρειαζόμαστε μόνο μία ΚΕΠΑ και μία κοινή εξωτερική δράση, χρειαζόμαστε και κοινή ενεργειακή πολιτική. Το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο επίσης θα εγκρίνει την πολιτική για τη Βαλτική θάλασσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την Επιτροπή και την Σουηδική Προεδρία που ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία. Το καθήκον του Συμβουλίου τώρα είναι να την εφαρμόσει αμελητή. Ελπίζω ότι η στρατηγική για τη Βαλτική θάλασσα θα τύχει της προσοχής που αξίζει από την Ισπανική και την Βελγική Προεδρία. Υποστηρίζω την ιδέα της Υπουργού Μάλμστρομ ότι θα μπορέσει να θεωρηθεί η στρατηγική της της ε, Βαλτικής ε, θάλασσας ως πρότυπο για άλλες ε, μακροπεριφερειακές πολιτικές. Αλλά δεν θα μας πάνουν στα σοβαρά αν δεν έχουμε επαρκείς πόρους για την εφαρμογή της πολιτικής. Η γραμμή του προϋπολογισμού χρειάζεται κονδύλια και αξιοπιστία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλα και τώρα κυρία Στρέλα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Μετά από το ναι στο δημοψήφισμα της Ιρλανδίας. Και μετά την τοποθέτηση του Πρόεδρου της Πολωνίας, ελπίζουμε ότι το, συντακτικό, το συνταγματικό δικαστήριο της ε, Δημοκρατίας της Τσεχίας θα δεχτεί τη συνθήκη και ο Πρόεδρος της Τσεχίας επίσης θα υπογράψει. Το Συμβούλιο δεν μπορεί να υποχωρήσει στην ε, εκβιασμό του Πρόεδρου τη Τσεχική Δημοκρατία. Η συνθήκη τη Λισαβόνα είναι άκρο αναγκαία για την καλύτερη λειτουργία των θεσμικών οργάνων τη Ευρώπη. Και έχει και άλλα πλέον εκτήματα. Συγκεκριμένα ενισχύει τι εξουσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα δικαιώματα των πολιτών. Έτσι είναι κατεπίγουσα η ανάγκη να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να θέσουν μια προθεσμία για τον πρόεδρο Κλάου, ώστε να συμπεριφερθεί ω πρόεδρο δημοκρατική χώρα μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αποδεκτό να σκεφτούμε καν ότι η βούληση ενός συγκεκριμένου κυβερνώντος μπορεί να αντιταχθεί στην βούληση της πλειοψηφίας. Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά τη Συνόδο της Κοπενχάγης. Ε, κύριοι και κυρίες, ο κόσμος μας χρειάζεται πραγματικά έναν πολύ σκληρό αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών, διότι έχουμε το φαινόμενο της θέρμανσης του πλανήτη που πλήττει, πλήττει και τις αναπτυγμένες χώρες και τις αναπτυσσόμενες. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να ενώσουμε τις προσπάθειές μας και να λάβουμε μια φιλόδοξη απόφαση. Η Κοπενχάγη είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε τις, να παραμποδίσουμε και να αναχαιτήσουμε την καταστροφή όπως μας προειδοποιούν οι επιστήμονες. Θα πρέπει λοιπόν να μην μειώσουμε τις φιλοδοξίες μας ε, στην ε, Κοπενχάγη. Η φιλοδοξία είναι απαραίτητη για να σώσουμε τον πλανήτη. Ευχαριστούμε κυρία Εστρέλα και τώρα για δύο λεπτά ο κύριος Μίτσελ. Um, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο πληθυσμό Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία γενιά θα αντιπροσωπεί 6% του παγκόσμιου πληθυσμού και δεν είμαστε πολύ πίσω τώρα. Οπότε δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή την εκπεριτροπή σε προεδρία ε, κάθε έξι μήνε ε, και να έχουμε πέντε διαφορετικά άτομα τουλάχιστον που θα μιλάνε για θέματα εξωτερική πολιτική εξονόμου τη Ένωση. Σε αυτή τη γενιά επίσης ο, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα έχει αυξηθεί κατά περίπου 2 δις. 90% ε, της αύξησης ε, θα παρατηρηθεί σε αναπτυσσόμενες χώρες 11, όπου 11 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο 5, 5 εκατομμύρια πεθαίνουν επειδή δεν υπάρχουν αρκετά ε, φάρμακα σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι μόνο σημαντικό να οργανωθούμε σε εσωτερικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να είμαστε εξοπλισμένοι, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε και τι καταστάσει στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Και γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι χρειαζόμαστε ισχύρη, έναν ισχυρό ανεξάρτητο επίτροπο για την αναπτυξιακή βοήθεια που θα έχει σαφή προπολογισμό και σαφή εντολή και θα είναι υπόλογο ή υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην αρμόδια επιτροπή. Είναι κέρια σημασία σε ύπατος εκπρόσωπο ή εν πάση περιπτώσει όποιο και αν είναι ο τίτλο του θα έχει ε, μεγάλο φόρτο εργασία, αλλά εδώ μιλάμε για ένα συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να υπερισχύει όλων, στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε. Δηλαδή, όχι μόνο πρέπει να μεριμνήσουμε τόσο ώστε να έχουμε έναν ισχυρό επιδίτροπο, αλλά αυτό το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να ανατεθεί σε κάποιον που θα αναλάβει σοβαρή δεσμεύση και έχει τα απαιτούμενα προσόντα, ούτω ώστε να ε, ε, αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Μίτσελ. Και τώρα για δύο λεπτά ο λόγος στην κυρία Μόνικα Μπένοβα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξότιμα Πρόεδρε του Συμβουλίου, κυρία Πίτροπε. Το πιο σημαντικό ζήτημα του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι κυρίως τη συνθήκη της Λισαβόνας και η διαδικασία εσωτερικής ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δρέωσής της στο διεθνές προσκήνιο. Θα πρέπει επίση να δούμε τα θέματα συνεργασία στον τρίτο πυλώνα, ε, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο αποτελεσματική, πιο δημοκρατική και πιο διαφανή. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να ασχοληθούμε με του βασικού ε, καρόνε των συνθηκών και την εσωτερική ενίσχυση τη ασφάλεια στην Ευρώπη. Εδώ χρειάζεται σεβασμό ε, των υπαρχόντων νομικών εργαλείων και ενίσχυση του επίση, λαμβάνοντα υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των πολιτών. Η ενίσχυση αυτών των δικαιωμάτων στον τομέα τη δικαιοσύνη και τη ελευθερία θα φέρουν πολλά πλέον πλεονεκτήματα σε όλου του πολίτε που θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στα δικαστήρια, τα εθνικά δικαστήρια και θα μπορούν να διασφαλίσουν τα δικαιώματά του και τι ελευθερίε του. Θα έχουν πλέον ελεύθερο δικαίωμα μετακίνηση και διαβίωση σε όλη την Ευρώπη. Η επιβολή του νόμου και η ενίσχυση τη ασφάλεια σε όλη την Ευρώπη είναι στρατηγική σημασία και πρέπει να αναπτυχθούν τέτοιοι στόχοι ώστε να αντιμετωπίσουμε αντιδράσει αντιδράσεις από κράτη-μέλη και από ανεύθυνους πολιτικού ηθήνοντε. Πρέπει να επιληθούν ευαίσθητα ζητήματα όπω η πολιτική μετανάστευση, του ασύλου ή τα ζητήματα των Ρώμα και άλλων εθνικών, εθνοτικών μειονοτήτων. Να μην μπορούν οι εξτρεμιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εκμεταλλευτούν τα θέματα αυτά. Έτσι λοιπόν η κύρωση τη συνθήκη τη Λισαβόνα θα είναι ένα πλεονέκτημα για όλου όσου τη υπογράψουν. Και η μεταναστευτική πολιτική τη Ευρώπη θα μπορεί να είναι και ένα κίνητρο για να ενισχύσουμε την αγορά εργασία των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχοντα υπόψη ότι θέλουμε αξιόπιστη και βιώσιμη πολιτική μετανάστευση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ζήτημα και τη λαθρομετανάστευση. Το οποίο για μα είναι σοβαρό πρόβλημα και για του πολίτε μα. Ευχαριστώ και τώρα το λέω και ο κύριο Μάουρο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Από καρδιάς, κύριε Πρόεδρε. Κουράγιο και πάλι κουράγιο. Αυτή είναι η δική μου σύσταση εν του επερχόμενου Συμβουλίου. Και αυτό γιατί θα συζητηθούν και οι διορισμοί των νέων επιτρόπων του Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ατόμων που μαζί με τον Πρόεδρο Μπαρόζο και τους υπόλοιπους επιτρόπους θα πρέπει να αναζωογονήσουν την ευρωπαϊκή πολιτική στο άμεσο μέλλον. Θα χρησιμοποιηθεί ω μέθοδο επιλογή αποκλειστικά το μέγιστο ωφέλιμα για του Ευρωπαίου πολίτε. Εδώ λοιπόν πρέπει να αναζητήσουμε άτομα με τέτοια πολιτική και ανθρώπινη υπόσταση που σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορούν να διακριθούν και να ασχοληθούν με τα κοινά ζητήματα που όλου μα απασχολούν. Αυτά θα πρέπει να είναι τα θεμέλια βάσει των οποίων θα συνεχίσουμε να μελετούμε σημαντικά ζητήματα όπως κλιματικές αλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εθνικών οικονομιών και την ε, οικονομική κρίση με την πρωτοβουλία, την ε, γενναία πρωτοβουλία του Eurobond. Και θα πρέπει αυτά να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Συμβουλίου. Συμπρασματικά να αναφέρω τα λόγια που ο Πάπας ε, είπε τα, τις προηγούμενες ημέρες εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Λόγια που θυμίζουν προληπτικά ότι έχουμε μια κοινή ευθύνη που αφορά όλους τους πολίτες, αλλά και όλους τους πολιτικούς ηθήνοντες. Ένα αίτημα να αναζητήσουμε την ένωση και την κοινή αναζήτηση της αλήθειας και να κάνουμε το αποφασιστικό βήμα για να οικοδομήσουμε κάτι σημαντικό για τους ίδιους τους αυτούς μας και τις ερχόμενες γενιές. ότι ο πρόοδος προέρχεται από τον πολιτισμό και η Ευρώπη βρίσκεται σε μία χρονική στιγμή που πρέπει να μεταδώσει τις αξίες που προέρχονται και από τον χριστιανισμό. Ε, το πολιτιστικό κληρονόμημα των λαών της Ευρώπης πρέπει να προβληθεί. Αυτό είναι ο δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τη σημαντική πρόκληση που έχουμε μπροστά μα, ώστε να ξαναγίνει πρωταγωνιστή στο κοινό προσκήνιο Ευρώπη. Ευχαριστούμε, κύριε Μάουρο. Και τώρα για δύο λεπτά η κυρία Ρόιτοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για μένα το βασικότερο σύστημα είναι η συνθήκη της Λισαβόνας ε, το τσεχικό συνταγματικό δικαστήριο ήταν συνεπές στις αποφάσεις και δεν νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα θεωρήσει ασύμβατη τη συνθήκη της Λισαβόνας με το τσεχικό ε, σύστημα. Ελπίζω εδώ να σταματήσει η τσεχική κόλληση ε, Ωστόσο η κυβέρνηση κάνει κατάχρηση εξουσίας. Δεν διορίζει ένα δικαστή στη θέση του επειδή χάσανε τη δίκη εναντίον του. Ναι, αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι. Δεν έχουμε θύμα ένα δικηγόρο ή ένα δικαστή, αλλά 500 ε, εκατομμύρια Ευρωπαίους. Και δεν έχουμε τις νέες εξουσίες, δεν μπορούμε να βγάλουμε κίτρινη κάρτα, κόκκινη κάρτα στα διάφορα θέματα, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη γρήπη, το έγκλημα, την τρομοκρατία, ε, να προχωρήσουμε σε ανθρωπιστική βοήθεια. Το ζήτημα που εκρεμεί, λέει, είναι η Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λόγω των διαταγμάτων ε, Μπενές. Ναι, μα αυτά είναι παράλογα πράγματα. Το άρθρο 345 της συνθήκης λέει ξεκάθαρα ότι ο χάρτης δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή. Ούτε ανοίγει νέο χώρο και διάστημα για αγωγές ε, σχετικά με ιδιοκτησίες. Και επίσης υπάρχει ένα νόμος το 2001 που ε, δεν μπορεί να ανατραπεί ε, και να επιστραφεί το, το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε μια κατάσταση που ίσχυε πριν από 50 χρόνια. Τι θέλει ο Κλάους. Θέλει τελικά να έχει την εικόνα ότι προστατεύει τις περιουσίες των Τσέχων από τους ξένους. Έχουμε αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα σήμερα ε, στη χώρα μας. Δείξτε λίγη υπομονή, θα το λύσουμε και μάλιστα πριν τις Βρετανικές εκλογές. Και θέλω να απευθύνω και μια έκκληση προς το Συμβούλιο ε, να υποστηρίξει την τσεχική ε, δημοκρατία στην προσπάθεια αυτή. Ευχαριστούμε τον κύριο Ρόιτοβα και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Παπαστάμκος για τη λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, η παρέμβασή μου θα επικεντρωθεί σε τρία σημεία. Σημείο πρώτο, η οικονομική κρίση. Η κρίση έπληξε αδιακρίτως όλα τα οικονομικά συστήματα ισχυρά και λιγότερο ισχυρά. η ανάγνωση της δεκάχρονης εμπειρίας της ονε υπό το φως της οικονομικής κρίσης καταδεικνύει την ανάγκη μεγαλύτερου ε, ρυθμιστικού εξευρωπαϊσμού της οικονομικής πολιτικής. καταδεικνύει επίσης την ανάγκη εξευρωπαϊσμού του οικονομικού κινδύνου. η εμπιστοσύνη είναι καλή ο έλεγχος είναι ακόμη καλύτερος σημείο δεύτερο κλιματική ε, αλλαγή. η ευρωπαϊκή ένωση ορθώς βρίσκεται στην πρωτοπορία της παγκόσμιας οικολογικής διπλωματίας. συμφωνώ απολύτως με το ε, ρηθέν υπό του προέδρου ε, Μπαρόσο, του προέδρου της κομισιόν ότι εν ώψη της διάσκεψης δεν υπάρχει σχέδιο β. κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το οικολογικό χρέος βαρύνει όλους ανεξαιρέτως. υποστηρίζω την ιδέα μιας παγκόσμιας τράπεζας κλίματος η οποία θα διαθέτει πόρους προερχομένους από το χρηματιστήριο ρήπων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η προσπάθεια των αναπτυσσομένων χωρών να αναπτύξουν να δημιουργήσουν ε, πρότυπα, αναπτυξιακά πρότυπα φιλικά προς το ε, περιβάλλον. Τρίτο σημείο είναι η μετανάστευση. Ασφαλώς πρέπει να προχωρήσουμε με ταχύτερους ρυθμούς στην καθιέρωση μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής. Όμως υπάρχουν και εξωτερικές πτυχές μετανάστευσης. Πρέπει να προχωρήσουμε τάχιστα στην εγκαθίδρυση αποτελεσματικών εξωτερικών σχέσεων με τρίτες χώρες ε, γιατί η πίεση προς τις χώρες ειδικά του Ευρωπαϊκού Νότου είναι μεγάλη. Ε, θέλω να πω ξεκάθαρα ότι η στάση της Τουρκίας είναι προκλητική. Χάρηκα που άκουσα ε, την Σουηδική Προεδρία να το επισημαίνει αυτό το μήνυμα της ευρωπαϊκής ένωσης προς την τουρκία αλλά και προς άλλες χώρες πρέπει να είναι σαφές ξεκάθαρο και αποτελεσματικό. αυτό το, πλαίσιο αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου και πρέπει να το σεβαστούν όλοι. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Παπαστάμκο. Και τώρα η τελευταία παρέμβαση από τον κατάλογο χωριτών. Ο κύριος Λίζε, για 1,5 λεπτό. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Σεσίλια Μάνστρομ και ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόσο αναφέρθηκαν στο κλίμα και την προετοιμασία της Κοπεχάκης και συμφωνώ με εκείνους που λένε ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει φιλόδοξα συμπεράσματα. Αλλά θέλω να σας προειδοποιήσω κιόλας και για τη χρηματοδότηση και για το ποιος θα κάνει τη μείωση τελικά και ποιος θα φτάσει στους στόχους. Πάντα Μιλάμε για την κλασική βιομηχανία που ε, ε, περιλαμβάνεται στο εμπόριο το 2005. Αλλά πάνω από 50% των εκπομπών ρήπων δεν ε, περιέχονται στο χρηματιστήριο των ρήπων. Χρειαζόμαστε περισσότερου ώμους για να σηκώσουν αυτό το βάρος. Ε, βλέπε ένα αέρια κυκλοφορία και βλέπε ένα αυσιπλοεία. Και μέχρι τώρα με έχουν απογοητεύσει και η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Εν ώψη του Πίτσμπουργκ, α πούμε, στο μέρασμα του Συμβουλίου δεν μπήκε αυτό το θέμα. Αν θέλουμε να πετύχει η Κοπενχάγη, τότε θα πρέπει να επιταχύνουμε, να πατήσουμε γκάζι. Τη Δευτέρα το έκανε η Επιτροπή περιβάλλοντο. Παρακαλώ να τα κοιτάξετε προσεκτικά αυτά τα δύο όλα θεσμικά όργανα. Το δεύτερο, ξέρω ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ άτυπο και μόνο, αλλά το Συμβούλιο σίγουρα θα μιλήσει και, και θα συζητήσει τη σύνθεση τη Νέα Επιτροπής, δεν μπορεί. Και με κάθε μετριοπάθεια θα ήθελα να προτείνω το εξή. Για λόγου ιστορικούς, ε, τα θέματα των φαρμάκων και το δίκαιο φαρμάκων ε, ήταν στη βιομηχανία. Και βέβαια τα φάρμακα είναι θέμα και τη φαρμακευτική βιομηχανία και το ε, αντίστοιχο δίκαιο, αλλά είναι και θέμα δημόσια υγεία. Αλλά ε, σε όλα τα κράτη-μέλη και στην Ένωση και ακόμα και στι Ηνωμένε Πολιτείε ε, είναι στο Υπουργείο Υγεία. Και θα παρακαλέσω να το εξετάσετε αυτό και να το διαβιβάσετε και στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιληφθεί λίγο αυτού του θέματος. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Λίζε. Και τώρα για δικασία κάτσε Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Λαντμπέργκης για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε του Συμβουλίου, ακριβώς εχθές εδώ ο κύριος Μπαρός, ο πρόεδρος, απάντησε ωραία στον κύριο Φαράτς και είπε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε τον πρόεδρο ε, του Συμβουλίου να είναι γνήσιος Ευρωπαίος. Είμαι βέβαιος ότι και οι σας και οι γύρω σας ε, αυτό το συμμερίζονται. Τώρα πρέπει να έχουμε ένα πραγματικό, ε, ένα γνήσιο γκασπρόμιαν, όπως είναι κάτι τύποι σαν το Σρόντερ, τον Πάβο Λίπονεν και τα λοιπά, ε, διότι της Γκάσπρομ. Και να τη φροντίζουν να έχουν καλές φιλικές σχέσεις και σχέσεις διαπλοκής και λαμογιάς και λαδόματος. Αυτός είναι ο δρόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι Ευρω... EU, είναι GU πλέον. Είμαστε η Ένωση της Gazprom έχουμε καταντήσει. Και θα πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση που η Ρωσία απολύτως αγνοεί πάντα την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δουλεύει ε, διαιρώντας την Ένωση. Παρακαλώ, τι λέτε εσείς, να βάλουμε κανέναν τύπο της Gazprom στην Προεδρία της Ένωσης. Ευχαριστώ να σας παρακαλέσω επίμονα και συγχωρήστε με αυτή την παράκληση, να περιορίζετε στο ένα λεπτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ αιτήσει για το λόγο. Να αφήσουμε όλου του συναδέλφου που θέλουν να εκφραστούν να το κάνουν. Να είστε λοιπόν περιορισμένοι στη διάρκεια τη παρέμβασή σα. Παρακαλώ. Το λόγο ζήτησε τώρα ο κύριος Γκάλαγκερ. Για ένα λεπτό. Δεν βρίσκεται στην αίθουσα. Η κυρία Γκάλαγκερ δεν είναι εντός εφούσης. Άριστα. Ο κύριος Πετρόσκη. Πρέγω. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η συνθήκη της Λισαβόνας ακόμη δεν έχει επικυρωθεί. Είναι ένα πολιτικό σχέδιο. Τι σημαίνει αυτό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη λαμβάνονται με ομοφωνία οι αποφάσεις. Όλοι μπορούν να ασκήσουν την ανησυχία και ο πρόεδρος Κλάους ε, δρά βάσει αυτών των κανόνων. Αν θέλετε να ασκήσετε πίεση σε αυτόν, τότε παραβαίνετε τους κανόνες, ε, γιατί ασκείται ουσιαστικά πίεση σε πολλούς πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακόμη αντιτίθεται σε αυτό το σχέδιο έχουν σοβαρούς ενδιασμούς. Έχουμε σύντομα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θεωρώ ότι οι πολιτικοί ηγέτες ε, θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το κατά πόσο αξίζει να παρακάμψουν την άποψη των πολιτών της Ένωσης. Ευχαριστούμε. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Τικάου, στην κυρία Τικάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει τη στρατηγική που αφορά την περιοχή της Βαλτικής θάλασσας. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι καλό μοντέλο για τη μελλοντική ευρωπαϊκή στρατηγική που αφορά την περιφέρεια του Δουνάβεως. Στην περιφέρεια αυτή τη Παραδουνάβια έχουμε 10 κράτη-μέλη, 10 κράτη, συγγνώμη, εκ των οποίων 6 ε, μέλη της Ένωσης και 200 εκατομμύρια ε, κατοίκους και το 75% ζει στις άμεσα βρεχόμενες από το Δούναβι περιοχές. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα πρόγραμμα δράσης, μια στρατηγική για το Δούναβι και μάλιστα πολιετές. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υιοθετήσουμε μέσα ε, χρηματοδοτικά για να αναπτύξουμε ε, οικονομίες αηφόρους και με αποδοτική χρήση ενέργειας και μιλώ εδώ για τις μεταφορές και για τα κτίρια. Το λόγο έχει ο κύριος Ζαν Ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε... κυρία Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ήθελα να ζητήσω από την κυρία Υπουργό, ίσως δεν με ακούει, να τη ρωτήσω μάλλον για την ε, εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Τη θέση σε ισχύ και την υπόσχεση ιδίω που έγινε μετά τον έτο τη Ιρλανδία ότι θα έχουμε έναν επίτροπο αναχώρα. Είχαμε κανονίσει το Δεκέμβριο του 2008 ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αναλάμβανε τα απαραίτητα νομικά μέτρα ώστε να έχουμε έναν επίτροπο τουλάχιστον αναχώρα. Κυρία Υπουργέ, ποια είναι αυτά τα νομικά μέτρα που θα ληφθούν. Ακούγεται η φήμη ότι θα τροποποιηθεί η συνθήκη τη Λισαβόνα με τη συνθήκη προσχώρηση τη Κροατία. Υπάρχουν και άλλε νομικέ διαδικασίε κατάλληλε Θα μπορούσατε να μα ενημερώσετε σχετικά με την είδηση αυτή που έφτασε σε εμά και πώ σκέφτεστε ο αριθμό των βουλευτών ε, με του 18 που θα έπρεπε να προσθεθούν στο νέο κοινοβούλιο με την Ευρωπαϊκή με την συνθήκη της Λισαβόνας. Πώς θα έρθει στο σωστό αριθμό αριθμό στο βουλευτό. αυτό. Ε, ευχαριστώ. Το λέω, κυρία Φιγκερέιδου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στο ερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα δοθεί άμεση προτεραιότητα στην μεταβολή των φιλελευθέρων πολιτών πολιτικών οι οποίε προκάλεσαν τη σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση. Χωρί ευαισθησίε και με τόλμη θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι συνθήκε φτώχεια, τι οποίε βρίσκονται τουλάχιστον 70 εκατομμύρια πολίτε ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τουλάχιστον 30 εκατομμύρια εργαζόμενοι με πολύ χαμηλού μισθού που δεν μπορούν καταφέρουν να ξεφύγουν από αυτό το επίπεδο φτώχεια διαβίωση. Θα πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να ε, αναζητήσουμε την απόκριση στη σοβαρή ανεργία που δεν σταματά να αυξάνεται και να μειώσουμε αυτά τα 30 εκατομμύρια στα ερχόμενα χρόνια. Θα πρέπει αμέσως να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα, τα μέτρα που απαιτούνται. Έτσι λοιπόν η μεγάλη πρόκληση για αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η ρήξη με τι φιλελεύθερε πολιτικέ, την ε, πολιτική τη Λισαβόνα και το Σύμφωνο Σταθερότητα. Θα πρέπει να κατασταθούν όλα αυτά από ένα πραγματικό πρόγραμμα κοινωνική και οικονομική πρόοδου, δίνοντα έμφαση στι ε, κοινέ υπηρεσίε τη ποιότητα, στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, στην αντιμετώπιση τη ανεργία και στην ε, ενίσχυση όσων εργάζονται, συμπεριλαμβανομένε τη ισότητα μεταξύ γυναικών και νέων. Ευχαριστούμε κυρία Φιγκερέιντο. Και τώρα ο κύριος Γκιωρή. Η κυρία Γκιωρή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καμιά φορά ορισμένοι θεωρούν ότι ε, θα πρέπει να σκεφτούμε ε, μήπως να αναγκάσουμε τον κύριο ε, Κλάους για να υπογράψει τη ε, συνθήκη της Λισαβόνας να εντάξει εκείνη και τα διατάγματα μπενές. Προσοχή, όχι, σας προειδοποιώ, αυτό είναι επικίνδυνο προηγούμενο γιατί ο κάθε ηθήνων στο εξή ε, θα μπορεί να θεωρεί ότι είναι σε θέση να επεμβαίνει στη συνθήκη και να την αλλάζει. Επικίνδυνο. Και η Σλοβακική κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ότι θα ακολουθήσει τη γραμμή του Κλάουσα αν περάσει. <coughs> Ιρλανδικό παράδειγμα. δεν ήταν νομικό το κόλλημα. Οι Ιρλανδοί ζήτησαν κάτι που υπήρχε στη συνθήκη και βγήκε. Επίσης, από τα 143 ε, διατάγματα Μπενές, 13 αφορούν ε, Γερμανούς και Ούγγρους και είναι άδικα. Ευχαριστούμε κυρία Ντατή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα συμφωνεί, θα, όπως και χτες, θα ήθελα να μιλήσω για την προετοιμασία της Συνόδου της Κοπενχάγης και για το ΕΚΟΦΗΝΕ που έγινε χτε και ουσιαστικά δεν εστέφθη με επιτυχία. Είχαμε ευθύνη ω βιομηχανοποιημένε χώρε να μεριμνήσουμε τόσο ώστε οι αναπτυσσόμενε χώρε να μπορέσουν να μα ακολουθήσουν στι προσπάθειες που κάνουμε για να καταπολεμήσουμε τι κλιματικέ αλλαγέ στην Κοπενχάγη. Μπορούμε να προσποιηθούμε ότι όλοι έχουμε τι ίδιε ικανότητε. Ε, γιατί, δηλαδή ότι όλοι ξεκινάμε από το ίδιο εφαλτήριο, αλλά δεν θα καταφέρουμε έτσι τίποτα οι εταίροι μα οι αναπτυσσόμενε χώρε για να μπορέσουν να μα ακολουθήσουν θα πρέπει να μην περιμένουν την ε, έκβαση του, τη Συνόδου της Κοπενχάγης. Θα πρέπει 27 να συμφωνήσουν οπωσδήποτε σχετικά με τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, δώσει την αναπτυξιακή βοήθεια λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές αλλαγές. Σας μίλησα για, για το ΕΚΟΦΗΝΕ που έγινε χτες. Ε, οι Υπουργοί Οικονομικών δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε κοινή θέση για αυτό το πρόβλημα παρά την κέρια σημασία του. η Επιτροπή με περιβάλλοντος ε, είχε κάνει σχετικές προτάσεις ε, και θα ήθελα να ε, μεριμνήσουμε τόσο ώστε να έχουμε την απαιτούμενη διεθνή αλληλεγγύη για να καταφέρουμε να ρυθμίσουμε αυτό το παγκόσμιο διάσταση πρόβλημα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκέρεντς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. θα απευθύνω ένα ερώτημα στην Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Ξέρετε ότι το βασικό πρόβλημα για, την για το μελλοντικό πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι αν αυτός ή αυτή θα ακολουθεί την κοινοτική μέθοδο ανεξαρτήτως των περιστάσεων. Θεωρείτε ότι αυτά τα κριτήρια πρέπει να είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για τον διορισμό του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εσχάτως ε, βλέπουμε μία διακρατική αποτυχία θα έπρεπε να θέσουμε τέρμα σε αυτή την περίοδο και να προάγουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να παραμείνουμε επίστη σε αυτό που οικοδόμησαν ε, οι κύριοι Μονέ και Σούμαν. Ευχαριστούμε κύριε Κεωρένς. Και τώρα το λόγο κυρία Αντζέλικα Βέρτμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, εμείς μιλάμε μόνο εντό εισαγωγικών το μόνο, για οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Γιατί δεν μιλάμε ποτέ για τη διορθωτική κρίση. Γιατί ξεκίνησε από μια πραγματική τραπεζική ε, κρίση στις επενδυτικές τράπεζες. Και μετά ε, παρασύρθηκε στη δίνη όλη αυτή και η υπόλοιπη οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Ρωμάνα Τζόρνταν Σιτζέλη. Ευχαριστώ. Ε, στις παραμονές της διάσκεψης Κοπενχάγη συζητάμε αυτά τα θέματα χωρί να έχουμε κάνει μεγάλα και πολλά βήματα από την προηγούμενη διάσκεψη. Δεν έχουμε μόνο τη χρηματοδότηση ω πρόβλημα, αλλά να δούμε πώς μπορούν να δεσμευθούν διάφορα κράτη και να τηρούν τις δεσμεύσεις τους ως προς τις εκπομπές ρήπων. Θα πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, διότι γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα εκεί έγκυται. Το Δεκέμβρη δεν θα θελήσουν και πάλι να αλλάξουν την ομοθεσία τους, αλλά εμείς θα πρέπει να το δονήσουμε. Και ήταν μεγάλη προεκλογική υπόσχεση του Ομπάμα αυτό ότι η Αμερική θα παίξει ρόλο ε, πρωτοποριακό και ε, προληπτικό στην καταπολέμηση αυτών των προβλημάτων. Και θα αξιοποιήσει, ελπίζω, ο Ομπάμα την ίδια του παρουσία εκεί για να πετύχει η διάσκεψη. Κόχλιτσεκ. κύριος Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, κυρία Επιτροπέ, συνάδελφοι. Σίγουρα το Συμβουλίο είναι ένα από τα βασικότερα θεσμικά μα όργανα και ασχολείται με θέματα και αρχών όπω πώ θα εξασφαλίσουμε θέσει εργασία και αξιοπρεπεί συνθήκε διαβίωση για του πολίτε μα. Εκπλήσω από δηλώσει πολιτικών κοινώντων που δείχνουν απόλυτη άγνοια των ζητημάτων αυτών. Και πολύ διαφορετικέ και αντικρουόμενες προσεγγίσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λοιπόν θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτές τις δηλώσεις και να φροντίσει να μην επικρατήσουν. Να λάβει μέτρα για την οικονομική ανάπτυξη και την βελτίωση της συνθηκών διαβίωσης των γεωργών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει την κοινωνική σφαίρα και τις ανάγκες των τραπεζών ώστε να μπορέσουν να πετύχουν μια θετική οικονομική ανάπτυξη στο μέλλον όσοι απελπισμένα θέλουν να, να, ήθελαν να παρεμποδίσουν το δημοψήφισμα για τη συνθήκη της Λισαβόνας, να τους θυμίσω ότι αν δεν μπορείτε να πενέψετε το σπίτι σας θα πέσει να σας πλακώσει. Και τώρα ο κύριος Δίας Ντεμέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μιλώ για τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε εσωτερικά και τη δικαιοσύνη. Πραγματική πολιτική μεταναστευτική ε, ενιαία ε, έλεγχος αποτελεσματικός των εξωτερικών συνόρων της ένταξης και του επανα, ε, επατρισμού. Eurojust και έλεγχος του Κοινοβουλίου. Αρμονική συνεργασία στη δικαιοσύνη, ποινική και αστική. Ε, λύση για το SWIFT, η δίκαια, προστασία των δεδομένων, προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και πολύ ισχυρή πρόθεση του χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων. Αυτά επιγραμματικά και ως κατάλογος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για τη συνθετική σας ικανότητα. Ο κύριος Γκέμπελς. Ευχαριστώ. Θα θέσω ένα πολύ απλό ερώτημα. Ε, θα διοριστεί διορίστηκε ο πρόεδρος μάλλον συγγνώμη της Επιτροπής, αλλά πότε θα έχουμε την Επιτροπή. Είναι αδύνατον να συνεχίσουμε με μια Επιτροπή όπου ε, πάνω από το ίμις των μελών ε, φτιάχνουν τα πράγματά τους για να φύγουν. Ε, χρειαζόμαστε σύντομα την Επιτροπή. Ε, Τώρα ο κύριος Λεπάσκορη. Η κυρία Λεπάσκορη. Δεν βρίσκεται στην αίθουσα. Η κυρία Λεπάς δεν είναι στην αίθουσα. Ο κύριος Κέλλη. Ε, I think one of the lessons to be learned... Νομίζω ότι ένα από τα μαθήματα που μπορούμε να κλείσουμε ποτέ κατά το δημοψήφισμα ε, τη Ιρλανδία ότι μια καλή εκστρατεία δημοσίων σχέσεων κάνει τη διαφορά. Τον Ιούνιο του 2009 ο Ιρλανδικό λαό ε, καταψήφισαν ε, μάλλον το 2008 καταψήφισαν τη συνδίκη της Λισαβόνας ε, και τώρα με δύο τρίτα πλειοψηφία την υπερψήφισαν. Έχει αλλάξει κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνυμα είναι ότι στάθηκε πολύ κοντύτερα τους η Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο ε, δημοψήφισμα. Ε, θα γίνουν καλά πράγματα υποσχέθηκαν, και, αλλά κυρίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε μια εκστρατεία δημοσίων σχέσεων για να πείσει τους πολίτες. Αλλά επί της ουσίας, ποια σχέδια έχετε ούτως ώστε ε, να διεξάγονται πιο ομαλά, αν θέλετε, τα δημοψηφίσματα στο μέλλον. Ευχαριστούμε. Η τελευταία παρέμβαση τώρα η κυρία, της κυρίας Λούναν. Ο, του κυρίου Λούναν. Βρίσκεται στην αίθουσα. Πρόεδρε, το όνομά μου είναι Λούχαν. Λούχαν. Κύριος ε, Λούχαν. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την διαδικασία κυρίωση τη συνθήκη τη Λισαβόνα, έχουμε ανάγκη τη συνθήκη αυτή για να λειτουργήσει σωστά η Ένωση και πρέπει να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη άμεσα η Τσεχία είναι το μόνο κατός που ακόμα δεν έχει κυρώσει τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θα πρέπει λοιπόν να απευθύνουμε έκκληση προς την Τσεχία ώστε ο πρόεδρος της, ο κ. Κλάους, να αναλάβει πλέον τις ευθύνες του και να κυρώσει τη συνθήκη πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο τέλος του μήνα Οκτωβρίου. Ιδάλλως θα βρεθούμε να μην μπορούμε να προχωρήσουμε τις θεσμικές μας συζητήσεις. Δεν θα μπορούμε να συγκεντρωθούμε στα πραγματικά προβλήματα, τις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Ευρώπης. Την οικονομική και δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, την ανεργία, την, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Δεν μπορούμε έτσι να διαμορφώσουμε και να σφυρατήσουμε την εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω πρωταγωνιστού στο διεθνέ προσκήνιο. Έχουμε μιλήσει διαμακρών για τι αρετέ τι συνθήκε αυτέ. Δεν πρέπει να παρατείνουμε άλλο αυτή τη συζήτηση. Αυτό που τώρα μα ενδιαφέρει είναι στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Επιτέλου να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία κύρωση τη συνθήκη. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν ολοκληρώσει. Πρέπει να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Δηλαδή να οριστεί η νέα επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λούχαν. Με συγχωρείτε για την κακή προφορά του ονόματό σα, του επιθέτου σα μάλλον. Τώρα η κυρία Μάλστρομ, εξ του Συμβουλίου, για να απαντήσει. Και μετά η Επίτροπος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους ε, βουλευτές για όλες τις ερωτήσεις τους ε, και τα σχόλια που έκανα. Μιλήσαμε πολύ για την Ευρώπη των πολιτών, των λαών και το ερμηνεύουμε ανάλογα με τους ιδίους ε, πολιτικούς στόχους. Εντάξει, δεν πειράζει, αλλά να ρωτήσουμε τους πολίτες τι θέλετε από την Ευρώπη σε όλες τις ευρωπαϊκές ε, χώρες ε, όλοι ζητούν ε, ευρωπαϊκή συνεργασία που βασίζεται σε κάποιες αξίες και ρυθμίζει τα κοινά μα προβλήματα. Η οικονομική κρίση δηλαδή, η ανεργία, οι κλιματικέ αλλαγές, η διασυνοριακή εγκληματικότητα, τα προβλήματα της μετανάστευσης κτλ. κτλ, κτλ. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Θα συζητήσουμε διάφορα θέματα σε δέκα μέρε ε, στη Σύνοδο Κορυφή. Ε, φυσικά δεν θα καταφέρουμε να τα ρυθμίσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον θα κάνουμε κάποια σημαντικά βήματα. Θα σημειωθεί πρόοδο ε, και ε, για να οικοδομήσουμε την Ευρώπη των πολιτών. Με δημοκρατικό τρόπο, με διαφάνεια πρέπει να λάβουμε τις αποφάσεις. Μπορεί να υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις για τις συνθήκες Λισαβόνας, αλλά η άποψη του Συμβουλίου και της Σουηδικής Προεδρίας και της πλειοψηφίας των βουλευτών ε, θεωρώ είναι ότι χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας θα προσεγγίζει περισσότερο τους πολίτες η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα λειτουργεί με πιο δημοκρατικό και αποτελεσματικό τρόπο και θα δώσει μεγαλύτερο ιδιαίτερο βάρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση παγκόσμια παγκόσμια σχέση τη. Γι' αυτό είναι σημαντικό να αρχίσει να ισχύει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, τόσο ώστε αμελητή να εφαρμοστεί η συνθήκη τη Λισαβόνα. Ακόμη έτοιμη λύση δεν έχουμε. Ούτε από την Τσεχική Προεδρία ε, Είχαν γίνει κάποιε προτάσει. Ε, θα συζητήσουμε με του φίλου μα στην Τσεχία για να βρούμε μία λύση και θα υποβάλουμε μία πρόταση για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά σα υπενθυμίζω ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο τη Τσεχία ε, οπωσδήποτε πρώτα πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση πριν μπορέσουμε εμεί να προχωρήσουμε. Ε, στο μεταξύ συνεχίζονται οι προετοιμασίε για τη συναπόφαση με το Κοινοβούλιο για την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση που θα συζητήσουμε το απόγευμα και θα επανέλθουμε σε πολλά από αυτά που υπόθηκαν σήμερα το το πρωί και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που σχετίζονται με τη συνθήκη της Λισαβόνα, Θα ε, συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Μπούζεκ για να δούμε πώς η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο μπορούν να συνεργαστούν ε, δυνάμει των νέων κανόνων. Μου έκαναν διάφορες ερωτήσεις για το Αφγανιστόν από τη Μαρία Ντεσένισε. Ναι, ελπίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση ε, για μια ευρωπαϊκή ομοθυμία για, το, για την πολιτική στο Αφγανιστάν, για την στρατιωτική παρουσία παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και μια αυξημένη στήριξη για την κοινωνία των πολιτών και για την ε, οικοδόμηση νέων υποδομών λοιπά. Θα δούμε πώς ακριβώς ε, θα στηρίξουμε και τις ε, νέες εκλογές που θα γίνουν σε 7 Νοεμβρίου και να στείλουμε παρατηρητές επιτόπου. Εν πάση περιπτώσει θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Ο μακροπρόθεσμος στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να έχουμε μια κοινή πολιτική ασύλου και μεταναστευτική μεταναστευτική πολιτική. Δεν θα το προλάβουμε μέχρι να αλλάξει ο χρόνο, γιατί χρειαζόμαστε τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίση, επεξεργαζόμαστε ακόμη το πρόγραμμα τη Στοχόλμη, ε, που ε, σχετίζεται και με τα μεταναστευτικά θέματα, που είναι ιδιαίτερα περίπλοκα. Μιλάμε για σχέσει με τρίτε χώρε, για το εμπόριο, ε, για την αναπτυξιακή βοήθεια για τη σύσταση νομικού πλαισίου για την νόμιμη μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αλληλεγγύη, για το σύστημα υποδοχής και θα υποβάλει αναφορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα βήματα που έχουν γίνει πριν ληφθούν περαιτέρω αποφάσει ε, το Δεκέμβριο. Τώρα για το πρωτόκολλο ε, της Βασιλείας. Είναι σημαντικό το θέμα. Λέμε συχνά ε, στους Τούρκους φίλους μας ότι θα πρέπει να το εγκρίνουν, να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν το πρωτόκολλο της Άγκυρες, αλλά δεν θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Θα συζητήσουμε τεθεί αυτό το θέμα το φθινόπωρο στις διαπραγματεύσεις ε, για την ε, ε, με την Τουρκία και θα ληφθούν αποφάσεις το Δεκέμβριο. Ε, αποφάσισε το Συμβούλιο ότι θα έχει κάθε χώρα έναν επίτροπο. Βάσει της ε, τωρινής συνθήκης ε, θα αλλάξει η κατάσταση το 2014. Μόλις τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε χρόνο για να δούμε ποιες νομικές προσαρμογές ε, πρέπει να κάνουμε ούτως ώστε να εγγυηθούμε ότι κάθε χώρα θα έχει το δικό της επίτροπο και θα πρέπει να συζητήσουμε με όλους τους νομικούς εθεσμούς ε, για να άτομα χρειάζονται τροποποιήσει ε, τη ε, συνθήκη ή αν επαρκεί μια ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου. Το ίδιο και για, τα 18, για τους 18 ε, πρόσθετους βουλευτές. Μόλις τεθεί σε ισχύ η συνθήκη θα αρχίσουν οι προετοιμασίες για την εφαρμογή και θα πρέπει να προετοιμαστούν τα κράτη-μέλη για να αποστείλουν αυτού του βουλευτέ εδώ στο Κοινοβούλιο και είναι περίπλοκο το θέμα των εθνικών εκλογικών συστημάτων. Θα χρειαστεί χρόνο. Ελπίζω να αρχίσουν οι προετοιμασίε το ταχύτερο δυνατόν. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που είπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι αυτοί οι βουλευτέ θα είναι παρατηρητέ στο μεταξύ έτσι, μέχρι να αναλάβουν επίσημα τα αξιώματά του και σε συνεργασία με την επερχόμενη Ισπανική Προεδρία θα μεριμνήσουν να καταβάλουν δυνατή προσπάθεια τόσο ώστε να είναι ομαλή η μετάβαση στο νέο σύστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το διάλογο. Ε, το Κοινοβούλιο προσφέρει μια ισχυρή στήριξη στην Προεδρία για τις κλιματικές αλλαγές. Ε, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο ώστε να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβει απόφασεις, για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δηλαδή την ευρωπαϊκή ε, συνεισφορά και τη δική μας συνεισφορά προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για να περάσουμε ένα ισχυρό μήνυμα στα πλαίσια των διεθνών διαπραγματεύσεων για να στεφθούν με μεγάλη επιτυχία ε, στην ε, Σύνοδο τη Κοπενχάγη. Είναι ένα σημαντικότατο θέμα για τη γενιά μα. Πρέπει να κάνουμε αυτά συγκεκριμένα βήματα για να καταπολεμήσουμε την αύξηση τη ε, θερμοκρασία και για να έχουμε ένα διεθνέ νομικό πλαίσιο. Σα ευχαριστώ για τη στηρίξη και για την αφοσίωσή σα και τη δέσμευση που δείχνετε σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Grazie, signora Malmström. Ευχαριστούμε κυρία Μάλστρομ. Και τώρα για την απάντηση και η Αντιπρόεδρος εκπρόσωπος της Επιτροπής, η κυρία Μάλστρομ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Μετά από αυτή την έντονη συζήτηση, ε, για την οποία σας ευχαριστώ, είναι σαφές ότι είναι κατεπίγουσα η θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτή η επιθυμία είναι χειροπιαστή πλέον και στη συζήτηση που έγινε και γενικά στο σώμα σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως και το Κοινοβούλιο είναι πρόθυμη και περιμένουν ανυπόμονα την θέση σε ισχύ της συνθήκης αυτής. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί λοιπόν η πολιτική διαδικασία που έχει ολοκληρωθεί στα περισσότερα κράτη-μέλη για την κύρωση και περιμένουμε από το κάθε κράτος μέλος να περατώσει τη διαδικασία κύρωσής του. Για να γίνει αυτό θα πρέπει βεβαίως να σεβαστούν τις εσωτερικές τους διαδικασίες. Βεβαίως, παράλληλα, είναι σαφές ότι κανένα επιμέρους κάτω μέλος δεν μπορεί να βρεθεί σε νομικό κενό. Οι αποφάσεις και οι καθυστερήσεις θα έχουν αντίκτυπο για όλους τους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν, είμαστε βέβαιοι ότι η Δημοκρατία της Τσεχίας πολύ σύντομα θα είναι σε θέση να κυρώσει τη συνθήκη και να θυμίσω σε όλους εδώ την ε, αγαστή συνεργασία που είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά και τα ιδιαιτερότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή που είχαμε πάντοτε ω τώρα. Είναι ζωτική λοιπόν σημασία τα κράτη-μέλη να εμπιστεύονται οι μεν δε ω προ τι δεσμεύσει που έχουν αναλυφθεί. Να σχολιάσω και το γεγονό ότι πολλά από τα μέλη του Κοινοβουλίου εδώ έχουν ε, κάνει μια σαφή διάκριση, ένα διαχωρισμό μεταξύ πραγματικότητας ανεργίας και οικονομικής κρίσης και του κειμένου της συνθήκης της Λισαβόνας. Ωστόσο, όλες οι ιδέες που ε, έχουν ε, προκύψει από τη συνθήκη της Λισαβόνας αφορούν ακριβώς το πλαίσιο. Θα είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι, με το οποίο θα μα επιτρέψει να είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι, να λάβουμε αποτελεσματικότερε αποφάσει και για τη μετανάστευση και για την πολιτική ασύλου, την ενεργειακή μα ασφάλεια, όλα όσα μα απασχολούν. Αυτό είναι ο στόχο. Θα πρέπει να διασυνδεθούν ε, όλα αυτά τα θέματα και θα είμαστε καλύτερα ε, προετοιμασμένοι για να τα αντιμετωπίσουμε. Και μετά θα περάσουμε και στη συζήτηση για τα θεσμικά ζητήματα. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα νέα αποτελεσματικά εργαλεία που μα προσφέρει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Η Επιτροπή λοιπόν εργάζεται εντατικά προετοιμαζόμενη για την υλοποίηση τη συνθήκη όταν τεθεί σε ισχύ. Σήμερα το απόγευμα γνωρίζω ότι θα ψηφίσετε θα ασχοληθείτε μάλλον και θα συζητείτε για την, με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Δεν είναι λοιπόν η στιγμή να περάσουμε τώρα στις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου ζητήματος. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω ότι εδώ υπάρχει μια σοβαρή πρόκληση. Πρόκληση να φέρουμε μαζί τους διαφορετικούς παράγοντες στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων και ο σφαιρικότερος στόχος μας, ο απότερος στόχος, θα είναι να καταλήξουμε σε διπλωματική συνεργασία. Έναν βαθμό δημιουργικής σκέψης θα τον χρειαστεί η εξέταση του θέματος αυτού. Επίσης πρέπει ταυτόχρονα να σεβαστούμε την διαθεσμική ισορροπία. Χρειαζόμαστε η υπηρεσία αυτή να έχει πλήρη υποχρέωση υπολόγου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι η δημιουργία ακριβώς της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης θα μας φέρει επιτυχίες αρκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστούν στενά. Πρέπει να σεβαστούμε ταυτόχρονα το γεγονός ότι ο ύπατος εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να κάνει κάποια πρόταση με τη σύμφωνη γνώμη τη υπόλοιπη Επιτροπής για ένα άλλο σημαντικό σημείο, επιτρέψτε μου να πω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε και η πρωτοβουλία για αυτού είναι κάτι που θα ξεκινήσει στα μέσα Οκτωβρίου με μια πράσινη βίβλο. Εδώ θα έχουμε ευρείε διαβουλεύσει με του πολίτε, ε, του εκπροσώπους τη κοινωνία των πολιτών και όλου του ενδιαφερόμενου για να ξεκινήσει σύντομα πρόταση ε, για, νομοθετικά κείμενα μετά τη θέση ισχύ τη συνθήκη οι επιπτώσεις της ε, χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης θα είναι από τις πρώτες προτεραιότητες των θεμάτων που θα εξετάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ακούσαμε πόσες αναφορές έγιναν στο θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της συζήτησης βεβαίως και συμφωνώ με όσους είπαν ότι δεν υπάρχει εδώ περιθώριο για συγκατάβαση η αδράνεια. Πρέπει να βρούμε πολιτική απόκριση στην κρίση και Ήδη βλέπουμε του πρώτου καρπού των προσπαθειών μα. Οι, οι χρηματοπιστωτικέ αγορέ αρχίζουν να εδρεώνονται, η εμπιστοσύνη αυξάνεται, όμω απέχουμε πολύ ακόμη από το να ανακάμψουμε πλήρω. Οι επιπτώσει στην απασχόληση είναι ορατέ και θα παραμείνουν, ε, παραμείνει οξύ το πρόβλημα. Οι πολιτικέ προσπάθειε λοιπόν πρέπει να συνεχιστούν, να εξακολουθήσουν για να στηρίξουμε την εργασιακή αγορά και τι πολιτικέ τη. Η Επιτροπή υποστηρίζει και το λέω αυτό απαντώντα σε κάποια από τα ερωτήματα που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια τη συζήτηση ε, υποστηρίζει τις προτάσεις για τον προπολογισμό και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο με την ψήφο του να επιβεβαιώσει αυτές τις φιλοδοξίες. Όπως είπε ο Πρόεδρος Μπαρόζο χθε, στη διάρκεια των ερωτήσεων, ως τώρα δεν έχουμε κάνει αρκετά, αυτό είναι σίγουρο. Η τωρινή κατάσταση είναι τέτοια που όλοι πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπαθίες μας και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Η ανεργία είναι σήμερα μία από τις πρώτες μας μέρημνες και ελπίζουμε πραγματικά να μας στηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπολογίζουμε σε εσά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Αλλά επίσης υπολογίζουμε σε εσά για να πιέσουμε το Συμβούλιο και σε εθνικό επίπεδο να πιέσουμε, ώστε να βελτιώσουμε ε, τις προτάσεις μας για την καλύτερη διαχείριση τα διαφορετικά ταμεία. Ένα άλλο ζήτημα που τέθηκε είναι αυτό του διοικητικού άχθους. Η Επιτροπή σύντομα θα εγκρίνει μία ανακοίνωση για τη μείωση του διοικητικού άχθους, η οποία θα ανακεφαλαιώνει όσες προσπάθειες έχουν γίνει ως τώρα, θα εντοπίζει ποια είναι τα βήματα που απομένει να γίνουν και θα αποφελείται από τις εργασίες της ομάδας Τρέντερ. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη αυτή ανακοίνωση, την έκθεση μάλλον, η εικόνα είναι γενικά θετική. Το διοικητικό άχθος και ο τρόπος να μειωθεί το διοικητικό άχθος βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο ω προ την εξέπρασή του. Οι περισσότερε προτάσει βέβαια εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου, οπότε και πάλι ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ασκήσει πίεση μαζί μα προ τα κράτη-μέλη, ώστε να αναλάβουν δράση και να προχωρήσουμε και στα ζητήματα αυτά. Επίσης να πω δύο λόγια για την ε, παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, την επίβλεψη. Αυτό είναι μια από, ένα από τα θέματα που βρέθηκαν στη μερίσια διάταξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανειλημμένω του τελευταίου μήνε. Ένα κατάλληλο ελεγκτικό πλαίσιο πρέπει να θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω ότι έχει επιτελεστεί σχετική πρόοδο. Υπάρχει ευρεία συνένεση σε επίπεδο Συμβουλίου για την πρόταση τη Επιτροπή για μακροοικονομική, ε, δομική και συστημική παρακολούθηση και έλεγχο, αλλά θα χρειαστούν πολύ περισσότερες προσπάθειες για την ε, μακροελεγκτική επίβλεψη. Θα πρέπει σύντομα να εξεύρουν μια φιλόδοξη και αποτελεσματική λύση. Επίσης, να πω και δύο λόγια για μια από τις πρώτες προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας, τις κλιματικές αλλαγές. Μένουν ακόμη λίγες εβδομάδες πριν από τη Σύνοδο της Κοπενχάγης και νομίζω ότι αρκετοί από εσάς έθιξαν το θέμα αυτό που θεωρούν ότι θα είναι το ζωτικό σημείο που θα καθορίσει το αν θα επιτύχουμε ή όχι. Χρειαζόμαστε κλιματική δικαιοσύνη, δηλαδή μια ισορροπία μεταξύ αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων χωρών. Το θέμα είναι πώς θα υποβάλουμε αξιόπιστες προτάσεις για τη χρηματοδότηση των μέτρων μετριασμού και προσαρμογής. Και θα πρέπει να αποδείξουμε την προθυμία μας να έχουμε εδώ ηγετικό ρόλο. Είμαστε οι μόνοι νομίζω που έχουμε υποβάλει πρόταση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χρηματοδότηση η οποία έχει γίνει αντικείμενο επίκριση από πολλούς ότι δεν είναι αρκετή. Σίγουρα δεν είναι αρκετή, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα. Είναι ένα πρώτο βήμα που αν όλα πάνε καλά θα κάνει και τους άλλους να εντατικοποιήσουν τι προσπάθειέ του, να προτείνουν και εκείνοι κάτι και όλοι μαζί να διαπραγματευτούμε στην Κοπενχάγη θα εξακολουθήσουμε να είμαστε δραστήριοι και δεν θα μειώσουμε το επίπεδο των φιλοδοξιών μας. Αντιθέτως, θα ενθαρρύνουμε όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και εταίρους να αναλάβουν πλήρως ε, τις ευθύνες τους, να καθίσουν γύρω μας το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, και να ασχοληθούμε με όλα τα προβλήματα και τις ανησυχίες των πολιτών. Σας διαβεβαιώ ότι δεν έχουμε την παραμικρή πρόθεση να μειώσουμε τις φιλοδοξίες μας. Αντιθέτως θα είμαστε δραστήριοι και ενεργοί ώστε να πετύχουμε μια καλή συμφωνία στην Κοπενχάγη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ την πρόεδρε Βάλστρομ. Κλείνει η συζήτηση. Σε δύο λεπτά θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Σας παρακαλώ λοιπόν να παραμείνετε στην αίθουσα, διότι εντός ολίγων λεπτών θα έρθει και ο Πρόεδρος για να ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες.